Guten Morgen. Καλή σας μέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί επισκέπτες, θα ήθελα να αρχίσουμε τη συνεδρίαση να σας χαιρετήσω αυτή την πρώτη α, συνεδρίαση του 2012. εγώ από απλώς για να μην εκπλαγείτε θα οργανώσω ε, τις εκλογές εδώ Προέδρου και Αντιπροέδρων γιατί είμαι η, ε, η βουλευτής η οποία έχει το περισσότερο η αρχαιότερη ας το πω έτσι βουλευτής εδώ της Επιτροπής λοιπόν βλέπω ότι είμαστε αρκετοί εδώ για να μπορέσουμε να κάνουμε τις εκλογές υπάρχουν ε, υπάρχει απαρτία δηλαδή. Αρχίζουμε λοιπόν με την εκλογή του νέου Προέδρου. Παρακαλώ προτάσεις, υποψηφιότητες. Ο κύριος Μπίλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να προτείνω τον κύριο Μάλκολ Χάρμπορ ως πρόεδρο της Επιτροπής δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνω εισαγωγή, να σας τον συστήσω. Είναι μέλος της Επιτροπής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ε, πραγματικά πιστεύει στην εσωτερική αγορά και τα δικαιώματα του καταναλωτή. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι εξαιρετικός πρόεδρος της Επιτροπής αυτής. Και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία αυτή για να τον ευχαριστήσω και όλα για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα στην Επιτροπή αυτή στο πρώτο ήμις Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπίλαν. Βλέπετε από το χειροκρότημα ότι είπατε τα σωστά λόγια. Άλλος που θα ήθελα να προτείνει άλλον υποψήφιο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν λοιπόν άλλες υποψηφιότητες. Οπότε ψηφίζουμε. Και μια και έχουμε έναν μόνο υποψήφιο, αν δεν υπάρχουν ενστάσεις να ψηφίσουμε διαβοής. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε. Ωραία λοιπόν. Ποιος είναι υπέρ του Μάλκομ Χάμπορ με της χειρός. Das ist einfach, eigentlich einfach fast alle πολύ εύκολο, σχεδόν ομοφωνία. Υπάρχουν κάποιοι που ψηφίζουν κατά, αποχές, όχι. Άρα λοιπόν, αγαπητέ Μάλκομ, εκλεγήκατε πρόεδρος ομόφωνα, χαίρομαι ιδιαίτερα. Καλή σας επιτυχία για τα επόμενα δυόμιση χρόνια. Σας παρακαλώ έρθετε εδώ να αναλάβετε την Προεδρία. <laughs> Uh, Κυρίες και κύριοι, μάλλον φίλοι και συνάδελφοι έπρεπε να πω, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την εμπιστοσύνη που επιδείξατε στο πρόσωπό μου και σας ευχαριστώ, ευχαριστώ ιδιαίτερα και την Μπάρμπαρα Βάιλερ που οργάνωσε την εκλογή αυτή και εκείνη έχει κάνει σοβαρή δουλειά και για το Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή ε, χαίρομαι που θα συνεργαστούμε και να λαμβάνω την προεδρία της ομάδας τώρα. Έχουμε ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα τους επόμενους 18 μήνες. Πάρα πολλά ε, θέματα πρέπει να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα και ο Πάνος Κωνσταντόπουλος θα μας βοηθήσει και σας ευχαριστώ που με υποστηρίξατε και ευχαριστώ επίσης και τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων που βρίσκονται εδώ. Ο φίλος Γιούργεν Κρόιτσμαν βρίσκεται ε, είναι ε, τώρα σε άλλη επιτροπή θα περιμένουμε να δούμε από τους φιλελεύθερους ποιος θα είναι ο, καινούργιο ο συντονιστής από εκεί και πέρα ε, έχουμε τον ε, τάτη του κυρίου Τριαντεφυλλίδη, ο οποίος έκανε επίσης πάρα πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια, αλλά ίσως θα έπρεπε να περιμένω να μιλήσω για τη δουλειά ε, την οποία πρέπει να κάνουμε και τον, να κάνουμε και τον απολογισμό της προηγούμενης ε, δουλειάς που έγινε εδώ στην Επιτροπή, στην Επιτροπή των Συντονισμών. Εγώ πάντως πιστεύω ότι η Επιτροπή μας κάνει πολύ σημαντική δουλειά και συνεχώς κερδίζει αξιοπιστία και αξία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζω επίσης και τους ακροατές γιατί η συνεδρίαση αυτή βγαίνει στο διαδίκτυο ε, και θα ήθελα να προχωρήσω στην εκλογή μάλλον πρέπει να κάνουμε και τις υπόλοιπες εκλογές που έχουμε να κάνουμε εδώ την προχωρώ στην εκλογή των αντιπρόεδρων τέσσερις ε, υποψηφιότητες υπάρχουν ε, που οι προτάσεις υπερβλήθησαν από τις πολιτικές ομάδες η κυρία Κόχαλε από το ΕΛΚ ο κύριος Τρεματέρα από το ΕΛΚ επίσης ο οποίος ασθενεί σήμερα γι' αυτό δεν είναι εδώ ο κύριος Γκρέκ από τους σοσιαλιστές και άλλος ένας υποψήφιος από τους σοσιαλιστές ε, αυτές οι προτάσεις υπερβλήθησαν από τις πολιτικές ομάδες δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες δεν υπάρχουν οπότε οι τέσσερις υποψήφοι εξελέγησαν και θα ήθελα να γίνει διαβοής η έγκριση η εκλογή των υποψηφίων αυτών θα ήθελα να ευχαριστήσω ο, τους υποψηφίους για την υποψηφιότητά τους και να καλέσω τους τρεις εξ αυτών που βρίσκονται στην αίθουσα να έρθουν στο βήμα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που οργανώσετε τόσο γρήγορα τη, τις ε, και, διεξήγατε τόσο γρήγορα τις εκλογές θα ήθελα εκ μέρους του κυρίου Τρεματέρα να ζητήσω συγγνώμη αλλά δεν μπορούσε να έρθει σήμερα στις συνεδρίες διότι όπως είπατε ασθενή Harbor ε, Ευχαριστώ πολύ έτσι κι αλλιώς έχουμε αρκετούς ε, αντιπρόεδρους εδώ οι οποίοι έχουν ε, αναλάβει, έχουν δουλέψει πολύ ήδη μέχρι στιγμή στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για το έργο τους αυτό και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία για τα επόμενα δυόμιση χρόνια. Πολύ καλά. Θα ήθελα τώρα να πω σε σχέση με το πρόγραμμα που έχουμε ε, για σήμερα. Έχουμε και κάποιες παρουσιάσεις για να ξεκινήσουμε καινούργια θέματα. Επίσης αύριο το απόγευμα έχουμε μια πολύ σημαντική ακρόαση την οποία, στην οποία θα ήθελα να σας καλέσω η, της κυρίας Γκέπχαρτ θα έρθουν και πάρα πολλοί ε, και για να μας μιλήσουν κατά τη διάρκεια αυτής της ακρόας. Θα ήθελα λοιπόν να συμμετάσχετε όσοι από εσά μπορείτε, όσο περισσότεροι μπορείτε και θα ήθελα επίσης να πω ότι έχουμε και μία εφημερίδα, ένα newsletter της Επιτροπής μας η οποία φαντάζομαι ότι σας μοιράστηκε ε, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκδότη και την Τζοάννα που είναι η κύρια ρεπόρτερ που για αυτή την εκδοσή, για αυτό το τεύχος έφτιαξαν ε, μία ε, αν θέλετε εορταστική εισαγωγή για το υπόλοιπο της θητείας ε, θα ήθελα να πω τώρα στους ακροατές μας ακούν από το διαδικτύο ότι μπορούν κάλλιστα να μπουν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής μας για να δουν το τεύχος αυτό του newsletter ε, το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι τα πρακτικά παλιότερων συνεδριάσεων η πρώτη είναι οι συνεδρίες του Αυγούστου θα ήθελα να τα ελέγξετε και αν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης μας αύριο βράδυ δεν υπάρχουν ενστάσεις τα θεωρούμε εγκεκριμένα το ίδιο και για τα υπόλοιπα πρακτικά Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Και προχωρώ τώρα στο πρώτο ουσιαστικό θέμα τη σημερινή ημερήσια διάταξη. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για να φτιάξουμε μια γνωμοδότηση, μια έκθεση ειδική ε, ε, πρωτοβουλία για την, μια πανευρωπαϊκή υπηρεσία e-call στα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη μετάδοση κλήσεων εκτέκτης ανάγκης από με βάση το 112 τηλεκλήσεις δηλαδή ε, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα αυτό εμένα προσωπικά διότι είχα κάνει πριν από 6-7 χρόνια στο Κοινοβούλιο αρκετή δουλειά για το θέμα αυτό. Δεν πρόκειται για καινούρια ιδέα και πραγματικά είναι εκνευριστικό το ότι έχει αργήσει τόσο πολύ να προωθηθεί το θέμα αυτό. Θα ήθελα να καλωσορίσω την εισηγήτρια, την κυρία Σένα Λοβά, η οποία βρίσκεται εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την θα δώσω βεβαίως το λόγο ε, και στους σκιώδεις εισηγητές ε, που είναι αρκετοί ε, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία και θα έχουμε μετά την ευκαιρία να συζητήσουμε την παρουσίαση θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Σεναλοβά Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, μετά την πολύ επιτυχημένη εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής μας, χαίρομαι διότι στο δεύτερο μισό της θητείας μας ξεκινούμε με μια έκθεση πάνω σε ένα θέμα το οποίο έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή του Ευρωπαίου πολίτη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποθεί πανελειμμένος ότι πράγματι ενδιαφέρεται για τα καθημερινά ζητήματα που αφορούν στον πολίτη. Θα έχουμε ένα πανευρωπαϊκό σύστημα λοιπόν επίγουσων κλήσεων. Έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το θέμα αυτό. Η θέσπιση του όλου συστήματος ήταν, κινήθηκε με πολύ αργούς ρυθμούς. Με εθελούσια βάση λειτουργούσε το σύστημα, αλλά δεν ήταν αυτό πολύ αποτελεσματικό. Θα μπορούσαν να σωθούν 2.500 άνθρωποι που βρίσκουν το θάνατο κάθε χρόνο. χωρίς λόγο. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό επιχείρημα το οποίο δεν πρέπει να λησμονούμε εξ αρχής, παρά τις δυσκολίες για την ε, εισαγωγή του συστήματος αυτού. Μας ενδιαφέρει η ασφάλεια στα οδικά δίκτυα, τα χαρακτηριστικά παθητικής ασφάλειας των αυτοκινήτων, τα οποία σχεδιάζονται έτσι ώστε να ελεγχιστοποιηθούν οι συνέπειες των ατυχημάτων. Ο συνάδελφος κ. Σκοκ στην ε, Επιτροπή για τις Μεταφορές παρουσίασε την έκθεση αυτή σχετικά με την οδηγία για τις μεταφορές και την ασφάλεια στους ευρωπαϊκούς δρόμους μέχρι το 2020. Έχει πολύ μεγάλο νόημα να πούμε ότι η δική μας ε, Επιτροπή είναι αρμόδια για το θέμα αυτό, διότι η δική μας Επιτροπή ασχολείται με τον τρόπο λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Δεν θα πρέπει η αγορά η ευρωπαϊκή να είναι κατακαιρματισμένη. Θέλουμε να έχουμε κοινά πρότυπα. Η κοινή εσωτερική αγορά να είναι κάτι το οποίο να ωφελεί όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι αποκλειστικές υπηρεσίες να με τα τραπούν σε υπηρεσίες προσβάσιμες σε όλους, αξιόπιστες και ασφαλείς. Ε, περί αυτού πρόκειται. Αυτό είναι η ηλεκτρονική κλίση. Θα ακούσουμε λοιπόν δύο παρουσιάσεις. Θα ακούσουμε τον κύριο Φάντεν Πάιλ από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος θα αναλύσει τις τεχνικές εξελίξεις των ε, προτύπων, των στάνταρ για την ηλεκτρονική κλίση. Και στη συνέχεια θα, ακούσουμε τον κύριο Ουρμπάνικ, Γενικό Διευθυντή από τη Τσεχία του, ε, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της σχετικής, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα θέματα ηλεκτρονικής κλήσης. Έχουν ένα δικό τους τέτοιο σύστημα στη χώρα αυτή και προχωρούν σε επιχειρήσεις διάσωσης με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι ένα σύστημα δηλαδή που έχει εφαρμοστεί <clears throat> εκεί επιτόπου και ήταν πολύ επιτυχημένο. Βασικό εμπόδιο είναι ότι δεν έχουμε στήριξη πανταχώθεν για ένα πανευρωπαϊκό σύστημα. Πρέπει να αναλύσουμε τις περιπλοκότητες και τις αμφιβολίες που νομίζουν κάποιοι ότι υπάρχουν στο σύστημα αυτό. Ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση να τα εξετάσουμε όλα αυτά τις επόμενες εβδομάδες. <coughs> Άλλωστε, Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες προσφέρουν στα αυτοκίνητά τους ε, τέτοιου είδους λύσεις, οι οποίες όμως κατά την άποψή μου θα πρέπει να λειτουργήσουν μόνο ως εναλλακτικές λύσεις. Θα πρέπει να θεσπιστεί και να εισαχθεί το σύστημα αυτό σε όλα τα οχήματα στην Ευρώπη. Το 70% των απαντώντων στις έρευνες επιθυμούν ε, την ενσωμάτωση τέτοιων συστημάτων ε, και δυνατοτήτων στα αυτοκίνητά τους, έτσι ώστε να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια. η ηλεκτρονική κλίση δεν θα πρέπει να προσφέρεται μόνο ως ε, ε, επιλογή στα αυτοκίνητα πολυτελείας, θα πρέπει να ενσωματωθεί, να είναι υποχρεωτική η δυνατότητα αυτή σε όλα τα ευρωπαϊκά οχήματα, τα οχήματα που κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Άλλωστε, ε, πάνω από το 40% των αυτοκινήτων είναι εξοπλισμένα με συστήματα ιδιωτικά έκτακτης κλίσης ή κλίσης εν γέννη σε ιδιωτικό πάντοτε επίπεδο. Όμως, να μπορεί κανείς να κάνει μια ηλεκτρονική κλίση και να αποσταλούν οι αρμόδιες διασωστικές δυνάμεις, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βεβαίως οι δυνάμεις διάσωσης θα πρέπει πάντοτε να ανήκουν στο δημόσιο τομέα και να μην αναλαμβάνεται αυτό το έργο από ιδιωτικούς φορείς. Πιστεύω ότι τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας είναι πολύ σημαντικά. Ε, προσδοκώ με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να συνεργαστώ με τους σκιώδεις εισηγητές και όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στη δουλειά αυτή. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ έχω δουλέψει πάνω σε αυτό το θέμα. Βλέπω ότι έχετε κάνει πολύ καλή έρευνα και είστε πολύ καλά καταρτισμένοι και κατατοπισμένοι. Έχουμε τον κύριο Τιερή Βαντερπίλ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο οποίος θα μας κάνει μια παρουσίαση για την κατάσταση με, υιοθετώντας την οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και περιμένουμε τον κύριο Ομπάνιεκ, Υπουργό Εσωτερικών της Τσεχίας, ο οποίος δυστυχώς έχει κολλήσει στην κίνηση και γι' αυτό έχει καθυστερήσει. Εάν ε, δεν έρθει εγκαίρος θα θέσουμε τις ε, ερωτήσεις εσάς κυρία εισηγήτρια και θα του τις μεταφέρετε. Κύριε Τιερή Βαντερπίλ, καλώ ήλθατε. Να πω στους διαδικτυακούς μας ακροατές ότι θα έχουμε και διαφάνειες στην αίθουσα, θα έχει, ότι μάλλον στο διαδίκτυο μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες, οι οποίες είναι πολύ κατατοπιστικές. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα Σα ευχαριστώ αγαπητά μέλη της Επιτροπής αυτής για την πρόσκληση που μου απευθύνεται να πάρω το λόγο σήμερα και να παρουσιάσω το Πανευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Κλήσης. Επιμένω στη λέξη πανευρωπαϊκός και το δεύτερο ε, μέρος της πρότασης είναι η λέξη δημόσια, δημόσια ηλεκτρονική κλίση. Δηλαδή βασίζουμε όλη την προσέγγισή μας στον τηλεφωνικό αριθμό 112. Εν συντομία να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε την παρουσίαση των διαφανειών. Ο Πρόεδρος, ναι, ε, προσπαθούμε να ε, φορτώσουμε το αρχείο για να το προβάλλει η οθόνη. Ε, δεν έχουμε προτζέκτορ αυτή τη στιγμή, αλλά μέσα σε όλα τα μέλη έχουν αντίγραφο επιχάρτου μπροστά τους και μπορούν να παρακολουθούν τις διαφάνειες. Πολύ καλά. Λοιπόν, να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί το σύστημα. Όταν σημειωθεί σύγκρουση οχήματος, το όχημα αυτομάτως θα αποστείλει, θα πραγματοποιήσει μία ηλεκτρονική κλίση 112 στον αριθμό 112 ανοίγοντας ένα διάβλο ε, επικοινωνίας ε, με, τη, με τα επίγοντα περιστατικά και θα μεταδώσει τα ελάχιστα στοιχεία που έχουν σχέση με το ατύχημα. Δηλαδή σε ποιο χρόνο, σε ποια τοποθεσία, ε, σε ποια οδηγική κατεύθυνση και άλλα σχετικά στοιχεία ε, για το, ε, για το ελόγο όχημα. Και κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να μεταδώσει και τον αριθμό των επιβαίνοντων. Δηλαδή, μπορεί να αναγνωρίσει τον αριθμό των επιβαίνοντων από τον αριθμό των ζωνών που έχουν ασφαλίσει. Τι περιμένουμε από αυτό το σύστημα λοιπόν, ότι θα σωθούν ζωές. Ήδη έχουμε ακούσει ότι περίπου 2.500 άνθρωποι ε, πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω απουσίας του συστήματος αυτού, θα μειωθούν και οι σωματικές βλάβες, οι τραυματισμοί κατά 10% διότι η... θα έρθει η βοήθεια γρηγορότερα από ό,τι θα ερχόταν με μία κλίση κινητής ε, τηλεφωνίας ή όποιας άλλης τηλεφωνίας. Και επίσης, διάφορες άλλες ε, οικονομικές επιπτώσεις θα μειωθούν και θα απαλληλθούν. Για παράδειγμα, αμέσως θα λάβουμε πληροφορίες για την ύπαρξη ατυχήματος, άρα η αστυνομία και οι ε, τροχονόμοι θα μπορέσουν καλύτερα να διοχετεύσουν την κίνηση και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και θα έχουν οι αρμόδιοι φορείς όλες τις πληροφορίες τις απαραίτητες για το ατύχημα πριν να φτάσουν καν επί τόπου επομένως θα μπορέσουν ήδη να προχωρήσουν σε παρακάμψεις ή θα μπορέσουν ήδη να ε, πράξουν τα δέοντα για να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες. Δηλαδή, ε, από τη στιγμή που εξ αρχής θα σταλούν οι πληροφορίες για το ποια μάρκα, ποιο αυτοκίνητο ποια μάρκας έχει υποστεί ατύχημα, αμέσως θα γνωρίζουμε ε, με ποιο ακριβώς τρόπο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον απεγκλωβισμό. Από εκεί και πέρα, η τεχνολογία αυτή υπάρχει από το 2003 περίπου. Ενίοτε έχουν προσφέρει αυτή την τεχνολογία επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Όμως το ποσοστό διείσδυσης στην αγορά παρέμεινε μικρό και τελικά για ε, λόγους που δεν έχουν να κάνουν με την ε, επιχείρηση και για λόγους κόστους συντήρησης ε, εγκαταλείφθηκαν αυτές οι λύσεις. Άλλωστε, κανείς ιδιώτης δεν μπορούσε να προσφέρει πανευρωπαϊκή κάλυψη στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπροσθέτως, θα έπρεπε, ή έπρεπε μάλλον, όλοι οι, όλες οι υπηρεσίες διάσωσης να μπορέσουν να λειτουργήσουν με πάνω σε διαφορετικές λύσεις που εδράζονται σε διαφορετικά πρωτόκολλα ε, επικοινωνίας. Και έτσι αυξάνονται τα κόστη που πρέπει να αναλάβει ε, αυτός ο φορέας. PSAP, ε, Private Safety Answering Points. Επομένως, τίθεται και θέμα κόστος. Τώρα, ως προς την ε, ε, αποδοχή από τους ε, χρήστες. Το Ευρωβαρόμετρο το 2006 έκανε αυτή τη μελέτη και το 2010 επαναλήφθηκε μια σχετική μελέτη και στις δύο αυτές μελέτες τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα. Άνω του 70% των απαντώντων ζήτησε την ενσωμάτωση του συστήματος αυτού, την υιοθέτηση δηλαδή. Και μετά τον έλεγχο σταθερότητας, το ESP, το οποίο ήδη έχει ενσωματωθεί στα αυτοκίνητα, είναι το δεύτερο πιο επιθυμητό χαρακτηριστικό από πλευράς χρηστών. Επομένως, είναι κάτι που ζητούν οι χρήστες που αποδέχονται, ε, να, ε, αποδέχονται ευρέως να υιοθετηθεί και να χρησιμοποιηθεί στα οχήματά τους. Εγώ είμαι μέλος μιας διεύθυνσης που έχει να κάνει με την έρευνα και βεβαίως πάντοτε η τεχνολογία ε, ορμάται από ένα ερευνητικό project στην αρχή. Είχαμε λοιπόν πάρα πολλές δράσεις έρευνας, κάναμε διάφορα πιλωτικά προγράμματα, πειράματα και είχαμε την ευκαιρία να εξάγουμε συμπεράσματα όχι μόνο για το εάν ε, μπορεί να υφίσταται μια τέτοια ε, τεχνολογία, αλλά και για το αν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους χρήστες. Έχουμε λάβει υπόψη μας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, είχαμε πάρα πολλές συσκέψεις ειδικών, εμπειρογνωμόνων, επιτόπου, παρουσιάσαμε τα δεδομένα σε όλες τις ε, συμμετέχουσες ε, μονάδες σε όλους τους φορείς και το πιο σημαντικό ε, που έχω να πω είναι ότι ανέκαθεν μπορέσαμε, μπορούσαμε να βασιστούμε στην ε, στεναρή στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οποία και σας ευχαριστώ θερμά. Το 2003 λοιπόν ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει τέσσερα ανακοινοθέντα αναφορικά με την ηλεκτρονική κλίση και την ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής. Το τελευταίο ανακοινοθέν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξεδόθη το 2009 και καταστούσε σαφές το, το εξής γεγονός. Εάν δεν, δεν υιοθετηθεί τελικά το σύστημα αυτό, η ηλεκτρονική κλίση στο 112, τότε ε, ίσως ενδεχομένως θα εξέταζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ενδεχόμενο να ε, προβεί στην υιοθέτηση κανονιστικών μέτρων. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε ξεκάθαρα ότι εάν δεν επαρκέσει η εθελούσια συμμετοχή, τότε θα αναγκαζόταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο ε, σκληρή προσέγγιση ε, πιέζοντας για την υιοθέτηση κανονιστικών ρυθμίσεων για το θέμα αυτό. Και στην αξιολόγηση αντικτύπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλησε τις ε, διάφορες επιλογές. Με την ιδιωτική ηλεκτρονική κλίση δεν ε, καλύφθηκε το σύνολο της αγοράς. Είχαμε χαμηλό ποσοστό διείσθησης μόνο στα αυτοκίνητα πολυτελείας και μόνο σε ορισμένες χώρες. Επομένως, η επιλογή ε, να ανατεθεί σε, στους ιδιώτες το σύστημα αυτό δεν λειτουργήσε. Η εθελούντια προσέγγιση της ηλεκτρονικής κλίσης το 112 με τα κοινά πρότυπα τα οποία ήδη έχουν καθοριστεί είναι η επιλογή υπαριθμών 2. Και έχουμε φτάσει στην εξή κατάσταση με αυτή την επιλογή. Ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας περιμένει τον άλλον να δράσει. Δηλαδή, ο φορέας τηλεπικοινωνιών περιμένει την εγκατάσταση του συστήματος από πλευράς αυτοκινητοβιομηχανίας οι υπηρεσίες διάσωσης, ε, αστυνομία, πυροσβεστική κλπ. Περιμένουν να εγκατασταθούν τα συστήματα στο όχημα, αλλά και να μπορούν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών να τους διαβιβάσουν τα δεδομένα πριν υιοθετήσουν οι ίδιες δημόσιες υπηρεσίες την, ε, να υιοθετήσουν ε, την εγκατάσταση δικού τους συστήματος τεχνολογίας και πληροφοριών για να μπορέσουν να δεχθούν τέτοιου είδους ηλεκτρονικές κλήσεις στον, στον στον αριθμό 112. Επομένως, ε, όλα αυτά μας οδηγούν στην επιλογή υπαριθμών 3, δηλαδή η υιοθέτηση κανονιστικών διατάξεων και ρυθμίσεων. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε οικονομίες κλίμακας. Οικονομίες κλίμακας και για την αυτοκινητοβιομηχανία και να έχουμε τελικά ε, θετική έκβαση, θετικό αποτέλεσμα στην, ε, στον λόγο κόστους ωφέλειας, ο οποίος αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στο 1,74. Επομένως, αυτή η τριμερής νομοθετική, νομοπαρασκευαστική μάλλον διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει με στόχο να καταστήσει ε, υποχρεωτική την εγκατάσταση ε, ηλεκτρονικής, εξοπλισμού ηλεκτρονικής κλήσης σε όλα τα καινούρια οχήματα και έτσι οι φορείς PSAP και οι φορείς τηλεπικοινωνιών να αναλάβουν τη διαχείριση των κλήσεων αυτών με βάση ε, τα κοινά πρότυπα και τον κανονισμό. Τα κοινά πρότυπα βεβαίω ε, είναι το προαπαιτούμενο. Στα αριστερά της διαφάνειας αυτής βλέπετε τι ακριβώς θα κάνετε. Δηλαδή ε, θα εγκρίνετε την υποχρεωτική εγκατάσταση ενός συστήματος μέσα στο όχημα, το οποίο θα βασίζεται στα πρότυπα ΣΕΝ Στη μέση της διαφάνειας ε, βλέπετε τον ρόλο των ε, φορέων κινητής τηλεφωνίας. Αυτό έχει ήδη υιοθετηθεί μέσω σύστασης. Να είναι σε θέση δηλαδή να λάβουν την ηλεκτρονική κλίση 112 και να την διαβιβάσουν, διαβιβάζοντας ε, το, την ελάχιστη ομάδα δεδομένων που θα πρέπει να σταλούν. Αυτό ήδη υπάρχει. Και στα δεξιά της οθόνης Βλέπετε τα κέντρα ε, επίγουσας ανταπόκρισης, άμεσης ανταπόκρισης στις επίγουσες, στις επίγουσες κλήσεις και ε, τον ρόλο που θα αναλάβουν στη συνέχεια. Είπα ήδη ότι έχουμε ήδη υιοθετήσει το Σεπτέμβριο του 2011 υιοθετήσαμε τη σχετική σύσταση για τους φορείς ε, κινητής τηλεφωνίας. Είναι ο κύκλος στη μέση στην προηγούμενη διαφάνεια. Επομένως το πρώτο κομμάτι ε, της κανονιστικής αυτής ρύθμισης ήδη υφίσταται. Με βάση τις συστάσεις αυτές θα πρέπει τα κράτη-μέλη να παράσχουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικών κλήσεων θα πρέπει να εργαστούν ε, στενά με τους φορείς διαχείρισης δικτύων ε, ώστε να εξευρεθεί ο καλύτερος, ε, η καλύτερη οδός δρομολόγησης όλων αυτών των κλίσεων. Τώρα, οι φορείς κινητής, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει ε, να είναι σε θέση να διαχειριστούν τις ηλεκτρονικές κλήσεις ακριβώς όπως ε, διαχειρίζονται τις άλλες κλήσεις στο 112. Δηλαδή οι κλήσεις αυτές παίρνουν προτεραιότητα εναντί όλων των υπολείπων και δεν χρεώνονται. Και θα πρέπει να ε, επισημάνουν ότι η κλίση αυτή είναι ηλεκτρονική κλίση και μάλιστα είναι κλίση που αφορά ένα συγκεκριμένο ατύχημα που έχει ήδη συμβεί. Η σύσταση βεβαίως είναι ένα είδος νομοθετικής ρύθμισης το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα σκληρό. Άλλωστε η Ένωση ε, των ε, φορέων GSM ήδη έχει δεσμευτεί στη υιοθέτηση αυτού του συστήματος και όλα αυτά είναι μέρος των ε, προαπαιτούμενων και των τεχνικών προδιαγραφών που θα υιοθετήσουν οι εταιρείε κινητής τηλεφωνίας στο μέλλον. Εάν η ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων δεν ε, είναι αρκετή, φανεί τελικά στο μέλλον δεν είναι αρκετή, ε, μπορούμε να υιοθετήσουμε ένα πιο σκληρό νομοθετικό ε, μέτρο βασιζόμενοι στην οδηγία για τις καθολικές υπηρεσίες. Τώρα, αυτή τη στιγμή ε, ποιο νομοθέτημα προετοιμάζουμε. Αυτά που έχουν να κάνουν με την εγκατάσταση μέσα στο όχημα του συστήματος αυτού. Στην ανακοίνωση του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το σύστημα ηλεκτρονικής κλίσης να εγκατασταθεί βάσει των προτύπων ΣΕΝ σε όλα τα αυτοκίνητα τύπου 1, δηλαδή επιβατικά, και ε, ε, στα μικρά φορτηγά μέσω της υιοθέτηση σχετικού κανονισμού. Και μετά την υιοθέτηση αυτού του κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από πλήρη διαβούλευση με τα σχετικά μέρη, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τους εμπειρογνωμόνες, θα ε, προσδιορίσει τους τεχνικούς κανόνες και τα τεχνικά προαπαιτούμενα. Πρώτα λοιπόν ο κανονισμός και μετά με πράξη κατεξουσιοδότηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει ε, τα, τις τεχνικές προδιαγραφές. Επομένως, αυτά είχαμε προβλέψει στην ανακοίνωσή μας το 2009 και αυτά δρομολογούμε αυτή τη στιγμή. Ο Πρόεδρος, ε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ε, επιταχύνετε λίγο για να μην καθυστερήσουμε. Λοιπόν, θα ολοκληρώσω την παρέμβασή μου με το PSAP. Πρόθεσή μας είναι να έχουμε μια πράξη κατεξουσιοδότηση, ούτως ώστε να ευθετηθούν οι προδιαγραφές ε, και η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, αν θέλετε, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Θα δώσουμε την εντολή στα PSAP να εγκαταστήσουν ένα σύστημα που θα μας επιτρέπει να λαμβάνουμε τις ηλεκτρονικές κλήσεις μαζί με τα ελάχιστα δεδομένα και πληροφορίες για το εν ατύχημα. Επομένως, όταν εγκριθούν αυτές οι ειδικέ προδιαγραφές, τι θα γίνεται τότε. Εάν θέλει ένα, κράτη, ένα κράτος μέλος να αναπτύξει αυτή τη δυνατότητα ηλεκτρονικής κλήσης, θα, θα πρέπει να συμμορφούνται με τις ειδικέ τεχνικές προδιαγραφές. Η υποχρεωτικότητα θα αρχίσει να ισχύει 12 μήνες μετά την υιοθέτηση των τεχνικών προδιαγραφών, όπου δει και μετά από ξελόγηση αντικτύπου. Το τελευταίο που θα ήθελα να σας δείξω είναι αυτό εδώ. Τα πρότυπα που έχουμε ε, χαράξει μαζί με το ΣΕΝ και το NSD. Προαπαιτούμενα για τη λειτουργία, μονάδα ανταπόκρισης για παράδειγμα, μπορεί, θα πρέπει να μπορεί κανείς να διαβιβάσει αυτή την κλίση και να διαβιβάσει τα δεδομένα μέσα σε τέσσερα δευτερόλεπτα. Πρωτόκολλα υψηλού επίπεδου που ε, υλοποιούνται και εφαρμόζονται στα συστήματα αυτά. Όλα αυτά τα έχουμε κάνει σε συνεργασία με τη ΣΕΝ και την ΕΤΣΙ και την, ε, ε, υιοθετώντας τα, το 3GPP δηλαδή ανοιχτά πρότυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον οποιονδήποτε. Και βεβαίως όλα αυτά συμπληρώνονται με μια πλατφόρμα εφαρμογής, υλοποίησης, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Και παρακολουθούμε την ανάπτυξη του συστήματος αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδελεχή αυτή παρουσίαση. Είχαμε χάσει την τελευταία διαφάνεια, αλλά επιβεβαίωσε αυτό που είπα προηγουμένω. Είναι ότι χρειάστηκαν 7 χρόνια για την ε, ανάπτυξη του θέματο αυτού και χαίρομαι ιδιαίτερα που στην Άλφος Δίτα Χόχα, που ήταν από του κύριου ηγητές στην Επιτροπή ε, Μεταφορών, ε, είναι παρόν. Θα έχετε την ευκαιρία λοιπόν να πάρετε σχετικά το λόγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ότι διαθετήσατε τη συνάντηση αυτή και μπορούμε να, μπορούμε να μιλήσουμε τη θεωρία αυτή στην πράξη. Το γενικό ε, η Επιτροπή Γενικού... Αυτή ήταν η πλέον εργαζόμενη πάνω στο θέμα αυτό. Χαίρομαι που είναι εδώ και η κυρία Μπάνα που θα μας δώσει και σχετικά μας, μας ετοίμασε και αυτές τις διαφάνειες. Ευχαριστώ και τον ε, κύριο Γιάννη Μπάνα από την Επιτροπή, από το Υπουργείο Ιστορικών που είστε ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος στην Επιτροπή μας σήμερα για να μας μιλήσετε σχετικά με την πρακτική σας εμπειρία της πιλωτικής εργασίας πάνω στην εφαρμογή της, ηλεκτρονικής, της ηλεκτρονικής κλήσης. Και ιδιαίτερα με αυτό το νέο που ακούσαμε σήμερα το πρωί, γιατί κάθε φορά μαθαίνουμε ένα νέο ακρονίμιο. Είναι το PSAP, δηλαδή τα σημεία κλήσης ε, δημόσιας ασφάλειας. Τα PSAPs. Θα το βρω κάπου που είναι εδώ πέρα. Public Safety Answering Points. Ε, αυτό, είναι, ε, αυτό μας δίνει το ακρονίμιο PSAP που είναι ουσιαστικά δηλαδή ε, σημεία απάντησης τηλεφωνικών κλήσεων για τη δημόσια ασφάλεια. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που είστε εδώ και σας δίνω το λόγο. Πατάτε το κουμπί δεξιά για να ανοίξετε το μικρόφωνο και έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ανάμεσά σας σήμερα. Είναι δεύτερη φορά που απευθύνομαι και ομιλώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, παρουσιάσω την οπτική της PSAP στα πλαίσια της εφαρμογής της ε, ηλεκτρονικής κλήσης. Αισθάνομαι ότι το PSAP, αυτά τα δημόσια σημεία κλήσης για την ε, δημόσια ασφάλεια, δεν είναι πάρα πολύ ισχυρά παρόν και δεν έχει πολύ δυνατή φωνή όπως θα έπρεπε. Περί πρόκειται. Αυτά τα σημεία, τα PSAPs, τα οποία υπάρχουν σήμερα και ασχολούνται και λαμβάνουν ε, κλήσεις κατεπήγοντος. Στην ε, Τσεχία έχουμε κάπου 15.000 τέτοιες κλήσεις κατεπήγοντος την ημέρα, στην Τσεχία. 15.000 κλήσεις λοιπόν που λαμβάνουν οι χειριστές, όχι απαραίτητα κλήσεις κατεπήγοντος, το 2011, έχω τα τελευταία στοιχεία εδώ, είχαμε 16.305 οδικά ατυχήματα ε, στα οποία παρενέβη η πυροσβεστική και η υπηρεσία διάσωσης, το οποίο σημαίνει λοιπόν ότι αυτά τα ατυχήματα ε, αντιμετωπίστηκαν από την υπηρεσία μας. Βλέπετε εδώ πέρα τον αριθμό. Αυτά τα σημεία απάντησης προφανώς αντιμετωπίζουν πρόβλημα σήμερα και τα προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει το πρόβλημα των ξένων γλωσσών και βέβαια υπάρχουν διακρατικές επιπτώσεις στην εφαρμογή του συστήματος αυτού και υπάρχουν επίσης και σιωπηλέ κλήσεις. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της ηλεκτρονικής κλήσης αλλά δεν είναι απλώς ο στόχος ε, της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών κλήσεων να λύσουν τα προβλήματα αυτά. Στη Δημοκρατία της Τσεχίας έχουμε ένα ποσοστό ε, περίπου 70% των ε, ψεύτικων, αν θέλετε, κλήσεων φάρσας. και χρειάζονται ουσιαστικά σε έξι δευτερόλεπτα να αποφασίσει κανείς τι θα κάνει. Προετοιμάζουμε νέα τεχνολογία λοιπόν στο NSAP που θα μας οδηγήσει σε πολύ σύντομο, συντομότερο χρόνο ε, των υπηρεσιών ε, αντιμετώπισης επιγόντων περιστατικών. Αλλά πρέπει να σμικρύνουμε και το χρόνο προτού η κλίση αυτή φτάσει τις υπηρεσίες ε, ε, διάσωσης και άμεσης παρέμβασης και θεωρούμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα είναι χρήσιμο. Στην Τσεχία ήδη λειτουργεί η σημαία ηλεκτρονικής κλήσης σε ενιαίο δίκτυο από τον ε, Αύγουστο του περασμένου έτους, από τον Αύγουστο του 2011. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσω της, εφαρμογής ενός πιλωτικού προγράμματος του HE Euro με εναρμονισμένες και διασυνδεδεμένες υπηρεσίες. Χρησιμοποιούμε δηλαδή έναν ιαίο αριθμό που φέρει το ειδικό σήμα, την, την σημαία δηλαδή ηλεκτρονικής κλήσης που μετα, μεταβιβάζει το κλήση στη δική μας υπηρεσία. Πρέπει να εναρμονίσουμε και να κάνουμε διαλειτουργικές τις διάφορες υπηρεσίες η ηλεκτρονική κλίση προφανώς στόχο έχει να σώσει ζωές. Σώζει λοιπόν ζωές μέσω της μείωσης του χρόνου επισκόπησης ε, του ατυχήματος με αυτοματοποιημένη ενεργοποίηση της κλίσης αυτής σε τέτοιες περιπτώσεις όπως αυτή που βλέπετε αυτού του είδους του οδικού ατυχήματος, μέσω παροχής καλύτερης πληροφόρησης σε ό,τι αφορά την τοποθεσία του ατυχήματος και ακριβή τοποθέτηση και παρέχοντας επίσης τεχνικές πληροφορίες σε σχέση με το αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι ο αριθμός VIN των vehicles, των διαφόρων αυτοκινήτων δηλαδή, που μας δίνει τη δυνατότητα να προετοιμαστούμε ανάλογα προτού φτάσουμε κιόλας στο σημείο ε, του ατυχήματος. Έχουμε αυτές τις διαφορετικές κάρτες για τα διαφορετικούς τύπους αυτοκινήτων και ο αριθμός VIN ε, μας δίνει προφορίες ό,τι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του αυτοκινήτου το οποίο έχει εμπλακεί στο ατύχημα. Επίσης, ε, σώζει ζωές ηλεκτρονική κλίση μέσω της ε, απλούστευσης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Η ηλεκτρονική κλίση, λοιπόν, στόχο έχει να απλοποιήσει και όλη τη διαδικασία και πρέπει να την κρατήσουν στο δυνατόν πιο απλή. Πρέπει να κάνουμε όσο δυνατόν λιγότερες αλλαγέ, ώστε να μην χάνουμε χρόνο και να μην δαπανούμε περιτά κονδύλια. Πρέπει να χρησιμοποιούμε χαρακτηριστικά τα οποία ήδη υπάρχουν στην αγορά, με τον τρόπο με τον οποίο είναι σχεδιασμένα, αλλά να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τις δυνατότητες που προσφέρουν. Μπορείτε να δείτε τώρα πώς είναι αυτό το, το σήμα ε, του ηλεκτρονικής κλήσης, την οποία χρησιμοποιούμε. Όταν ε, εμφανίζεται στην οθόνη οποιοδήποτε κινητού ο αριθμός 112, δρομολογείται μέσα στο δίκτυο με τα πλέον κατάλληλο σημείο PSAP, την πλέον κατάλληλα διτοποθεσία του σημείου απάντησης δημόσιας απάντησης της ασφάλειας. Όταν θα εμφανίζεται και θα ενεργοποιείται το σήμα της ηλεκτρονικής κλήσης, το δίκτυο θα δρομολογεί διαφορετικά την κλήση αυτή, είτε στο κέντρο του PSAP, λήψης είτε μέσω άλλου σημείου εισόδου για την κλίση που θα είναι εξοπλισμένο με την κατάλληλη τεχνολογία για την αναγνώριση του αυτοκινήτου κλπ. Και η κλίση θα σηματοδοτείται συγκεκριμένα και ιδιαίτερα για τον χειριστή της, ε, του σημείου λήψης της κλίσης. Χρειάζεται όλοι να λειτουργούμε και να μην βρίσκουμε εμπόδια και να είμαστε αποφασισμένοι ότι θα λάβει χώρα. Γιατί ουσιαστικά όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει. Εφαρμόσαμε ένα πιλωτικό σχέδιο στην Τσεχία το 2007 και αυτό ήταν στην πρώιμη φάση ενεργοποίησης του συστήματος, αλλά ήδη προσπαθούμε να ελέγξουμε τις διάφορες προδιαγραφές για να δούμε πώς θα λειτουργούν στην πραγματικότητα. Οφείλω να πω ότι κατεβλήθη πάρα πολλή δουλειά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οργανισμούς τυποποίησης και θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό ε, την ευκαιρία εδώ τους οργανισμούς αυτούς. Σήμερα έχουμε ολοκληρώσει με το κομμάτι των προδιαγραφών και ελέγχονται σε πιλωτικά προγράμματα. Βλέπουμε ότι οι προδιαγραφές λειτουργούν σωστά. Και η ιδέα η αρχική ήταν σωστή. Και... As good for us is uh, delays. The delays which are caused by... Ορισμένες φορές ε, είναι, υπάρχουν ε, αντίθετες αλλαγές ό,τι αφορά διαφορετικά στοιχεία. Για παράδειγμα, υπάρχει, υπάρχει ένα πεδίο αναλογικού τύπου σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Για τις υπηρεσίες απλοποίησης, αυτό δεν είναι κάτι σημαντικό, γιατί έχουμε το ίδιο αυτοκίνητο τον ίδιο τύπο αυτοκινήτου να λειτουργεί είτε με βενζίνη, είτε με πετρέλαιο, είτε με φυσικό αέριο, υγροποιημένο αέριο. Και αυτό για μας δεν αποτελεί καμία διαφορά σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές του αυτοκινήτου. Αλλά στα πλαίσια της κλίσης η οποία έρχεται προκαλεί προκαλεί πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία τυποποίησης. Από την άλλη, υπήρχε ένα πεδίο αντιμετώπισης σε ό,τι αφορά τις, ε, την προσφορά των διαφόρων προμηθευτών, σε ό,τι αφορά ε, το σημείο αυτό, αλλά πλέον δεν υπάρχει. Αυτό το οποίο πρέπει πραγματικά να κάνουμε και είναι υποχρεωτικό στην ηλεκτρονική κλίση είναι να ξέρουμε ακριβώς πού θα απευθυνόμαστε στις πιο τεχνικής υφής προφορίες, αυτές τις προφορίες που δεν έχουμε σήμερα. Αυτές οι αλλαγές λοιπόν, οι πληροφορίες που δεν είναι χρήσιμες, θα πρέπει ε, να αναγνωριστούν και να εξαιρεθούν. Αυτό που λέω πάντα στην όλη πλατφόρμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις διάφορους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι ότι πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση και ενιοποίηση όλων αυτών των αλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο δημόσιος τομέας στα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να δαπανίσει χρήματα εάν ε, η εισαγωγή αυτού του συστήματος δεν αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση. Θα ήθελα να, να, να, συγκρίνω αυτή την πλατφόρμα της ηλεκτρονικής κλήσης με τη σχετική υπηρεσία για την βοήθεια των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η ηλεκτρονική κλήση θέτει υποχρέωση στα κράτη-μέλη που θα διασφαλίζει ότι τα άτομα με κινητικές δυσκολίες και με ειδικέ ανάγκες θα έχουν ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, όπως και ένας απόλυτα φυσιολογικός πολίτης. Όμως δεν υπάρχουν ε, πρότυπα για κάτι τέτοιο. Από την άλλη, έχουμε ένα τεράστιο κατάλογο προτύπων για την ηλεκτρονική κλίση, αλλά δεν έχει επιβληθεί καμία υποχρέωση στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν το σύστημα προς το παρόν. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να δουλέψουμε στο πεδίο της ε, πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο θέμα, γιατί οτιδήποτε επενδύσουμε, πιθανόπατα θα αλλάξει με κάποια νομοθετική πράξη Ευρωπαϊκής Ένωσης του χρόνου ή σε δύο χρόνια. Και επομένως θα, τα κονδύλια θα πάνε χαμένα. Γι' αυτό και δεν επενδύουμε στο σημείο αυτό. Ξέρουμε ότι έχουμε υποχρέωση, αλλά πρέπει να υπάρξει προηγούμενη τυποποίηση. το αποτέλεσμα του έργου αυτού, του ευρωπαϊκού project, το οποίο έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών της ε, Τσεχίας, που είναι υπεύθυνο για την ε, καθολική εφαρμογή της ε, οδηγίας σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφορικής. Μπορείτε να δείτε την εικόνα αυτή, μια εκδοχή δηλαδή της ηλεκτρονικής κλίσης. Στο μέσον υπάρχει πλήρης πληροφόρηση σε ό,τι αφορά τις ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται να δοθούν. Και αυτό είναι το, εικόνα που πώς θα, του πώς θα φαίνεται, αν θέλετε, η, το αρχείο πληροφόρηση μέσω μιας ηλεκτρονικής κλήσης. Είχα την ε, τιμή να, να παρουσιάσω στην ε, κυρία Σενάλογα την ε, εικόνα αυτή και καταφέραμε να, να δούμε πειραματικά, πιλωτικά, αν θέλετε, την πραγματική λειτουργία της ηλεκτρονικής κλήσης, πώς μεταδίδεται και πώς μεταβιβάζεται μέχρι την υπηρεσία κατεπήγοντος πραγματικά λειτουργούσε το σύστημα και δεν ε, φοβάμαι να πω ότι λειτουργεί το σύστημα ηλεκτρονικής κλήσης στην Τσεχία. Το θέμα είναι να ενσωματώσουμε αυτή την εκδοχή στο πραγματικό σύστημα των PSAP. Οι πληροφορίες επίσης παρουσιάζονται στο χάρτη μέσω των συντεταγμένων, των γεωγραφικών συντεταγμένων του ατυχήματος, βλέπετε το άνισμα της ταχύτητας, οπότε ο χειριστής έχει την πλήρη πληροφόρηση σε ό,τι αφορά την διεύθυνση, την, τοποθεσία, την ακριβή τοποθεσία του ατυχήματος, το άνισμα της φοράς και όλα αυτά καθιστούν την διαδικασία λήψης απόφασης πάρα πολύ σύντομη. Βλέπετε την ακριβή τοποθέτηση μέσω της ηλεκτρονικής κλήσης από πού έχει γίνει, οπότε μπορείς να στείλεις το πυροσβεστικό επιτόπο. Καταληκτήρια λοιπόν συμπεράσματα. Εάν αυτή η εφαρμογή ήταν εφικτή το 2007, σίγουρα θα είναι πολύ πιο εφικτή και να εφαρμοστεί στις μέρες μας με καλύτερη τυποποίηση και καλύτερες τεχνολογίες. Και στο τέλος του Project Hero που προβλέπεται το 2013 θα έχουμε πλήρη, ε, πλήρωση επιχειρησιακή την ηλεκτρονική κλίση για την Τσεχία, ε, έτοιμο το σύστημα για οποιοδήποτε ε, όχημα με τυποποιημένο πανευρωπαϊκό όμπου και προσκαλώ οποιοδήποτε άτομο στην αίθουσα να το δοκιμάσει. Ελάτε στην Τσεχία και δοκιμάστε μόνοι σας το σύστημα ηλεκτρονικής κλήσης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Uh, well, thank you very much indeed. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και μας κάνετε την παρουσίασή σας. Χαίρομαι που από τη μια είχαμε μια παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την άλλη μεριά είδαμε πώς εφαρμόζονται ορισμένα πράγματα σε ε, συγκεκριμένη χώρα. Ε, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Σενάλοβα για να μας πει πώς τι πώς θα ήθελε να προωθηθεί αν θέλετε αυτό το θέμα γιατί μιλάμε για έκθεση ιδίας πρωτοβουλία την οποία θέλουμε να προωθήσουμε αλλά ίσως πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια να δώσω το λόγο σε άλλους που ίσως θα ήθελαν παρέμβουν ε, και οι σκιώδεις συγητές είναι εδώ και ο κύριος Δεγιόγκ και εγώ και ο κύριος Σάβη και η κυρία Ράπτη βεβαίως η οποία ήταν η συγγήτρια για την έκθεση Δίας πρωτοβουλία για το 112 ε, υπάρχουν και η κυρία Γκέπχαρτ και πάρα πολλοί άλλοι που έχουν ασχοληθεί με συναφή θέματα λοιπόν θα σας δώσω το λόγο αλλά εστέλα κονική παρακαλώ διότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας Λοιπόν, για να δω τώρα. α αρχίσω με την κυρία Ράπτη, η οποία ήταν η προηγούμενη εισηγήτρια για να μα πει τι έχει γίνει μέχρι τι έγινε. Και μετά θα προχωρήσουμε στου κοιόδες εισηγητέ, την κυρία Τούν, Ντε Γιόγκ, εγώ, Πέντεργαστ, Βανιού, Πουζόη και Γκέπαρτ. Η κυρία Ράπτη. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια. Είμαι πολύ ευτυχής που συνεχίζετε να είστε πρόεδρος αυτής της Επιτροπής. Σας εύχομαι καλή δουλειά. Ε, να πω ότι συνήθως γκρινιάζω όταν είναι εδώ η Επιτροπή και μιλάει. Αυτή τη φορά δεν θα γκρινιάξω, θα πω συγχαρητήρια στην Επιτροπή. Ε, είπε εξαιρετικά πράγματα, αισθάνομαι ότι προχωράμε και αυτό με ευχαριστεί γιατί είναι για το καλό των Ευρωπαίων πολιτών. Το τρίτο σημείο είναι ότι όταν άκουσα για εκείνο το PSAP, ξέρετε εγώ είμαι από την Ελλάδα όπου συζητάμε συνεχώς για το PSI. Μόλις άκουσα λοιπόν PSAP η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει, λέω φτάσαμε μέχρι εδώ, χρειαζόμαστε το 112 για να σωθεί η Ελλάδα. Ε, κάνω λίγο χιούμορ γιατί καταλαβαίνετε ότι βοηθάει σε αυτές τις στιγμές. Ε, θέλω να πω ένα ακόμη ευχαριστώ στην Εύελιν Γκέπχαρτ, την συντονίστρια των σοσιαλιστών, που μου έκανε τη τιμή να είμαι εισηγήτρια στο ψήφισμα για το 112. Ένα ψήφισμα το οποίο ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούλιο στο Στρασβούργο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία και επίσης θέλω να πω ένα ευχαριστώ στην συνάδελφο Όλγα Σενάλοβα διότι αισθάνομαι ότι η δουλειά από μένα μετά πέρασε σε ακόμα καλύτερα χέρια κάνει εξαιρετική δουλειά. Ε, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι το 112 πρέπει να ζήσει, πρέπει να εξαπλωθεί και πρέπει να είναι στη ζωή μας για να έχουμε τη ζωή μας. Ε, μία ερώτηση θα κάνω στον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ε, το κόστος. Πόσο θα κοστίσει από τη μεριά των κρατών μελών. Νομίζω ότι σε αυτούς τους καιρούς της οικονομικής κρίσης που περνάει η Ευρώπη είναι σημαντικό το κόστος, θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και θα πρέπει ανάλογα να πορευτούμε έχοντας στο μυαλό μας πάντα ότι πρέπει να σώζουμε ζωές. Ευχαριστώ και πάλι. Um, okay. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν να προχωρήσουμε στους σκιώδες, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κόχ. Ήταν εισηγητής στην Επιτροπή Μεταφορών και, και για εισηγητής για θέματα οδικής ασφάλειας. Οπότε ε, θα θέλαμε να ακούσουμε ε, μερικά σχόλια από την οπτική γωνία της Επιτροπής Μεταφορών. Κύριος Κόχ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα το απόγευμα θα ε, συζητήσουμε πάλι το θέμα στην Επιτροπή Μεταφορών για να δούμε πώς μπορούμε κι εμείς να εμπλακούμε. Αλλά ε, θα, τώρα δεν θα συμφωνήσω με την προλαλή σας, διότι εγώ απογοητεύτηκα λιγάκι από αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί μιλάει για στάνταρτ, για πρότυπα, για διάφορα πράγματα, για την εισαγωγή της ηλεκτρονικής κλήσης. Ωραία, αλλά αυτά είναι ιστορία δεν μας είπε τίποτα καινούριο. Δεν άκουσα να γίνονται τα βήματα εκείνα προόδου τα οποία θα επιθυμούσα να ακούσω. Περίμενα να μας πει η Επιτροπή από την τάδε ημερομηνία είναι υποχρεωτικό σε όλα τα οχήματα να ισχύει, να υπάρχει εγκατεστημένο το σύστημα της ηλεκτρονικής κρίσης. Τίποτα από αυτά δεν είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επανέλαβε ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να γίνουν τα επιβατηγά και τα μικρά φορτηγά και για τα άλλα οχήματα. Κρίμα ε, λοιπόν ε, λέω εγώ από πλευράς μου απογοητεύτηκα ζητούμε ξανά σα, και, και εγώ και εκ μέρους της Επιτροπής Μεταφορών να γίνουν τα λόγια πράξεις κάτι αυτό πρέπει να κάνουμε πια Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι. Και επειδή είπατε ότι θα συνεργαστείτε και μαζί μας, ε, αν υπομονούμε να συνεργαστούμε με την Επιτροπή, Μεταφορών. Κυρία Τούν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που πήραν το λόγο σήμερα. Φαίνεται ότι επαναλαμβάνουμε βέβαια όλοι ότι η ασφάλεια των πολιτών μας, των ε, ε, οδηγών, των επιβατών είναι πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό είναι προφανές ε, και βεβαίως προσπαθούμε να μειώσουμε και τα τροχαία ατυχήματα. Αυτό όλοι θέλουμε να το κάνουμε, αλλά πολλά πράγματα παραμένουν ακόμη ασαφή. Θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε κάπως τη δουλειά μας και να την επιταχύνουμε. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στο 112. Δεν λειτουργεί σε ολόκληρη την Ευρώπη όπως θα έπρεπε το νούμερο αυτό γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια αναφερόμαστε στις ηλεκτρονικές κλήσεις και πάλι δεν έχουν οριστεί ημερομηνίε, δεν έχουν οριστεί συγκεκριμένα projects ενώ όλοι πιστεύουμε ότι το θέμα έχει έναν επίγοντα χαρακτήρα και θα έπρεπε να προωθηθεί γρήγορα. Η Επιτροπή Μεταφορών ε, ε, εργάζεται και αυτή για το θέμα αυτό αλλά θα πρέπει και αυτή να ε, επιταχύνει το έργο της ε, και να υπάρχει πολλά ακόμα, πολλή ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει. Ο επόμενος ομιλητής λέει ο πρόεδρος είναι ο κύριος De αν και δεν ξέρω ποιος είναι ο σκιώδης από τους πράσινους. Θα δώσω το λόγο στον κύριο De μετά έχουμε Pendergast και και διάφορους άλλους ομιλητές Γι' αυτό έστε παρακαλώ σύντομη, γιατί πρέπει να κάνουμε, έχουμε και μια ψηφοφορία που πρέπει να κάνουμε ακόμη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ πρώτα πρώτα για την εκλογή σας στην Προεδρία της Επιτροπής. Δεν ξέρω αν θυμάστε... Ε, ε, Παλιότερα ε, μιλούσαμε για τα μεγάλα, τις μεγάλες πολιτικές ομάδες που αναλαμβάνουν όλες τις προεδρίες. Εσείς είστε από μια μικρότερη ομάδα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Λοιπόν, για το θέμα που συζητούμε, έχω ασχοληθεί με το ε, κα, 112 ως νούμερο ε, έκτακτης ανάγκης ε, είναι κρίμα που δεν μπορούμε ακόμη να εξηγήσουμε στους πολίτες της Ευρώπης ότι αυτό το 112 δεν είναι το ενιαίο νούμερο σε ολόκληρη την Ευρώπη και ότι μπορεί να, σε κάποιες χώρες να, να πρέπει να χρησιμοποιήσουν άλλα νούμερα είναι κρίμα πρέπει να επιταχύνουμε τη δουλειά μας Λοιπόν, εδώ μιλάμε για ένα καινούριο σύστημα το οποίο θα εγκατασταθεί σε όλα τα οχήματα υπάρχει μεγάλο ποσοστό κλήσεων φαρσών όπως αναφέρθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο στην Τσεχία φαντάζομαι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει προβλέψει μηχανισμούς αποφυγής αυτών των κλήσεων εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τώρα συγκεκριμένα πόσο θα ανέβουν οι τιμές των αυτοκινήτων εάν γίνει το σύστημα αυτό υποχρεωτικό για όλα τα αυτοκίνητα και θα ήθελα να αναφερθώ τώρα και στην παρουσίαση του κυρίου Ουρμπάνεκ. Καταλαβαίνω ότι ενοχλείται που δεν έχουν εφαρμοστεί ορισμένα πράγματα ακόμη. Α, είπε ότι χρειάζονται αλλαγές ποιες αλλαγές, όχι σε πρότυπα φαντάζομαι, αλλά σε τεχνικές προδιαγραφές, ποιες είναι αυτές οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Μπορεί να μας πει μερικά παραπάνω πράγματα και ίσως θα έπρεπε να ακούσουμε από τα διάφορα κράτη-μέλη που δεν έχουν εφαρμόσει το σύστημα αυτό και συμφωνώ με την κυρία Ράπτη, μάλλον απηχώ το ερώτημά της, ότι πρέπει να μας πείτε πόσο θα κοστίσει το σύστημα αυτό για τα κράτη-μέλη. Ε αλλά γενικώ είμαι υπέρ του συστήματος προφανώς. Ε, πρόεδρος, ευχαριστώ για τα ερωτήματα. Ε, ίσως δεν πάρουμε απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα σήμερα, αλλά τα σημειώνουμε και φαντάζομαι ότι θα απαντηθούν ίσως αργότερα. Η κυρία Πέντεργκάρστ είναι η επόμενη ομιλήτρια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε και θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ για την εκλογή σου ως πρόεδρο της Επιτροπής αυτής. Ε, επανεκλογή μάλλον. Ε, χαίρομαι που θα συνεχίσεις το έργο σου. Στα μέσα της προηγούμενης χρονιάς 22 κράτη-μέλη είχαν ε, συμμετάσχει στο σύστημα που συζητούμε. Αυτή τη στιγμή ποια είναι η κατάσταση θα θέλω να ρωτήσω και γιατί υπάρχουν κράτη που δεν συνυπέγραψαν αν θέλετε την πρωτοβουλία αυτή. Πολύ καλή, πολύ καλή ερώτηση λέει ο πρόεδρος, δυστυχώς η δική μου η πατρίδα είναι αυτή που δεν έχει συν συν υπογράψει. Κυρία Γκέπχαρτη επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις που έγιναν και να αναφερθώ σε κάτι που είπε ο κύριος Σουρμπάνεκ. Ο κύριος Σουρμπάνεκ είπε ότι δεν πρέπει να ζητούμε τα πάντα ή να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πάντα. Είναι σωστό αυτό και θα ήθελα να το, τονίσω και, να το τονίσω κι εγώ. Εδώ πρόκειται για την ασφάλεια των πολιτών μας, για την υγεία τους, για τη ζωή τους. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ο νίος μέχρι ότου να γίνει κάτι τι. Θα πρέπει να φροντίσουμε να ξεκινήσει το σύστημα να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε και να πούμε έστω ότι ξεκινούμε ένα σύστημα το οποίο δεν είναι ακόμη τέλειο, αλλά αρχίζουμε να το εφαρμόζουμε και θα το βελτιώσουμε μέχρι ότου να είναι τέλειο. Αν περιμένουμε από την αρχή να είναι τέλειο το σύστημα, θα περιμένουμε ονείως φοβάμαι. Αυτό θα ήθελα να το τονίσω. Ευχαριστώ πολύ ο Κρίστιαν Ιουζόη, ο ομιλητή, πολύ σκιώδη συγητής, ε, πολύ ενεργό σκιώδη συγητή για τις καθολικέ υπηρεσίες. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε η συνάδελφός μου κυρία Περβάνοβα είναι η σκιώδη συγγήτρια εγώ παίρνω το λόγο σήμερα για να, πάρω να πω τρία πράγματα πρώτον ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι υπάρχοι υπηρεσιών κινητής ε, τηλεφωνίας θα συμμετάσχουν ε, στο νούμερο αυτό το 112. Δεύτερο θέμα, υποστηρίζω στεναρά τη σύσταση που λέει ότι όλα τα κράτη-μέλη να φροντίσουν όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών τους για την κινητή πληροφορία για την κινητή τηλεφωνία συγγνώμη, να συμμετάσχουν στη ε, διαχείριση αυτή των κλήσεων 112 για να τους δώσουν προτεραιότητα. Τρίτο θέμα, θα πρέπει όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας να εγκαταστήσουν συστήματα που θα εντοπίζουν τις κλήσεις 112. Δεν είναι επιπλέον κόστος αυτό, είναι επένδυση που θα σώσει ζωές. Πρέπει να γίνει. Η κυρία Βανιού. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη γιατί δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ελέγχθηκαν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σενάλοβα και τους άλλους που πήραν το λόγο για τις προφορίες που μας έδωσαν. Θα ήθελα και εγώ να κάνω έκκληση όπως και οι άλλοι συνάδελφοι έκκληση να προχωρήσουμε. Εδώ και τέσσερα χρόνια δουλεύουμε για τα θέματα καθολικών υπηρεσιών είχαμε πει ότι το 112 είναι απαραίτητο απαραίτητο το νούμερο αυτό για την ασφάλεια των πολιτών η Κομισιόν το Κοινοβούλιο θα πρέπει να φροντίσουν, να υποκινήσουν τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν με τους ε, παρόχους κινητής τηλεφωνίας για να ξεκινήσει το σύστημα. Θα μπορούσαμε πράγματι να τελειοποιήσουμε αργότερα το σύστημα, αλλά ας αρχίσουμε να το λειτουργούμε τώρα. Πρέπει να υπάρξει η πολιτική βούληση για να ξεκινήσει το σύστημα πανταχού στην ε, Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Είναι προφανές, μπορούμε να το κάνουμε. Απλά πρέπει να συμφωνήσουμε και να ξεκινήσουμε τη λειτουργία του. Όλοι μαζί. Ο κύριος Άριας... Παρακαλώ πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Θα ήθελα να θέσω επιτάπητο στο εξής. Ποιες φόρμουλες, αν θέλετε, χρησιμοποιεί αυτό το μοντέλο επίγουσων κλίσεων για να διαβιβάσει πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος. Υπάρχει επικοινωνία μεταξύ ε, του κέντρου επικοινωνίας και του επιβαίνοντα. Με, σε τι γλώσσα θα μιλήσουν. 27 γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η αρχική γλώσσα στην οποία ε, θα διαβιβαστούν οι πληροφορίες για το ατύχημα αυτά. Για παράδειγμα, όταν νοικιάζει κανείς ένα αυτοκίνητο. Νοικιάζει κανείς ένα αυτοκίνητο σε μια άλλη χώρα από τη δική του και παθαίνει ένα ατύχημα. Πώς θα με επικοινωνήσει και σε ποια γλώσσα θα μιλήσει. Πώς θα λυθούν όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Uh, right. well, um... Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε στις ψηφοφορίες, αλλά έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Κύριε Βαντεπίλ, πολλά τα ερωτήματα, δεν μπορείτε να τα απαντήσετε όλα σήμερα. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο για το χρονοδιάγραμμα. για το ποια θα είναι η φύση της νομοθετικής αυτής πρότασης. Όλα αυτά θα ήταν χρήσιμα για την Επιτροπή μας. Και μετά, ε, κύριε Ορμπάνεκ, θα δώσω και σε εσά το λόγο για να κάνετε τα καταληκτικά σχόλια. Ο κύριος Βαντερπίλ, στα πρώτα απ' όλα, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι Στηρίζετε όλοι θέρμο το 112 και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Αυτή η στήριξη στο 112 και στην ηλεκτρονική κλίση είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα, ως προς την, ε, το χρονικό πλαίσιο. Στόχος μας είναι το 2015 όλα τα οχήματα να είναι εξοπλισμένα με αυτό το σύστημα ηλεκτρονικής κλίσης, επιβατικά οχήματα και ελαφρά φορτηγά. Κατηγορίας 2. Τώρα το κόστος. Κόστος ανάπτυξης για τα οχήματα θα γίνουν οικονομίες κλίμακα στα υφιστάμενα οχήματα, εν πάση περιπτώσει 80 ευρώ αναόχημα. Αυτό υπολογίζουμε. Και για το PSAP Πολύ μικρό είναι το επιπρόσθετο κόστος από τη στιγμή που ήδη έχουν εγκαταστήσει το σύστημα για να δεχθούν τις κλήσεις 112. Μεταξύ 30.000 και 300.000 ευρώ αναλόγως με το μέγεθος του εκάστοτε φορέα, δηλαδή της εκάστοτε μονάδας ανταπόκρισης σε επίγουσες κλήσεις για θέματα δημόσιας ασφάλειας. Public Safety Answering Point. Τα δεδομένα διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς και ε, είναι στη γλώσσα ε, του φορέα. Ένα γαλλικό αυτοκίνητο, ας πούμε, ταξιδεύει στην Αγγλία. Θα, ε, δι, θα λάβουν οι υπηρεσίες δεδομένα μεταφρασμένα στα αγγλικά από τη στιγμή που το ατύχημα συμβαίνει στην Αγγλία. Τώρα, για την επικοινωνία μεταξύ του φορέα και του αυτοκινήτου, ναι, ανοίγει μία δίωδος φωνής, αν θέλετε, δεδομένων φωνής, ή ε, μπορούν να την ανοίξουν χειρονακτικά οι επιβαίνοντες στο όχημα. Τώρα, ως προς τον αριθμό των προσώπων. Είναι μία πληροφορία που διαβάζεται αυτομάτως. Γιατί ε, μετράει ο αισθητήρα πόσες ζώνες έχουν δεθεί και άρα ε, από εκεί εξάγει την ε, πληροφορία για το πώς οι επιβαίνοντες βρίσκονται στο όχημα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Να δώσω το λόγο και στον κύριο Ορμπάνεκ για να κάνει κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις αν το επιθυμεί. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις άκουσα και θα ήθελα ε, να παρατηρήσω το εξής. Το κόστος για, το, για τους PSAP. Δεν μπορώ να παρουσιάσω ένα νούμερο. Δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Ωστόσο, το κόστος της εφαρμογής της υλοποίησης του συστήματος της ηλεκτρονικής κλήσης εξαρτάται βεβαίως από μια τεχνολογία η οποία ήδη χρησιμοποιείται στο κράτος μέλος. Αν το κράτος μέλος έχει εξοπλιστεί με τη σύγχρονη τεχνολογία PSAP, το κόστος, ε, το επιπρόσθετο της συμπερίληψης της ηλεκτρονικής κλήσης δεν είναι καθόλου υψηλό. Είναι καλή τιμή δηλαδή για αυτό το οποίο παίρνουμε. Αν τώρα το κράτος μέλος έχει την παλιά τεχνολογία, η οποία δεν δίνει αυτή τη δυνατότητα, δεν παρέχει καλές υπηρεσίες, τότε Μιλούμε γενικότερα ε, για το ότι το σύστημα 112 θα χωλένει στο εν λόγω κράτο μέλο που έχει την παλιά τεχνολογία. Επομένω, αναγκαστικά το κράτο μέλο θα πρέπει να επενδύσει παραπάνω. Αλλά όχι λόγω της ηλεκτρονικής κλίσης, Λόγω του ότι πρέπει να αναβαθμίσει την υπηρεσία 112 που γενικότερα προσφέρει στους πολίτε του. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, η γλώσσα, ο γλωσσικός φραγμός. Όπως είπα στην παρουσίασή μου, όντως τίθεται αυτό το θέμα στο 112. Το 5% των κλήσεων γίνονται σε ξένη γλώσσα. Και ε, αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να λύσουμε και πριν την ε, θεσμοθέτηση της ε, ηλεκτρονικής κλήσης. Δεν υπάρχει τρόπος να ξέρουμε ποια γλώσσα θα μιλάει ο οδηγός μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ένα αυστριακό τηλέφωνο, να κάνει μια ηλεκτρονική κλίση και να μιλήσει ιταλικά. Από τα στοιχεία που λαμβάνουμε δεν μπορούμε φυσικά να γνωρίζουμε ε, ποια γλώσσα θα μιλήσει ο επιβαίνων στο όχημα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι πρόβλημα του συστήματος ηλεκτρονικής κλήσης αυτό. Τίθεται με πρόβλημα, αλλά πρέπει να λυθεί σε άλλο επίπεδο, της γενικότερης πρόσβασης στις ε, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, στα επίγοντα. δεν θα πρέπει αυτοί οι δύο λόγοι να καθυστερήσουν ε, τη διαδικασία, γιατί δεν άπτονται αμυγός της ε, ηλεκτρονικής κλήσης. Σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ. Έχετε εμπειρία στην πράξη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι, ήμουν σκιώδης εισηγητής, δεν μίλησα εγώ καθόλου για το θέμα αυτό, όμως τα στοιχεία που μας δείξατε ε, είναι ξεκάθαρα και δεν έχουν καμία σχέση με τη γλώσσα. Άλλωστε, όταν συμβαίνουν σοβαρά ατυχήματα, οι υπηρεσίε σα ε, θα έχουν πολύ περισσότερα στοιχεία και πληροφορίε από ό,τι είχαν στο παρελθόν για το συγκεκριμένο ατύχημα που συμβαίνει, ε, ανεξαρτήτως γλώσσα. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικό όφελο, ε, το οποίο ε, δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί. Κυρία Σαναλόβα, να σα δώσω το λόγο να είστε σύντομοι, παρακαλώ, για να προχωρήσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αδράξω αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε για να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν, ε, όλους όσους έκαναν σχόλια. Συζητήσαμε τα τεχνικά ζητήματα, είδαμε την εμπειρία που υπάρχει στην πράξη και είδαμε βεβαίως από τα σχόλιά σας ότι υπάρχει και πολιτική βούληση για την ε, εγκατάσταση των ε, συστημάτων αυτών. Πριν ε, ε, τη σύνταξη αυτής της έκθεσης θα συσκεφθώ με τους σκιώδεις εισηγητές να δούμε όλες τις πτυχές του ζητήματος, να δούμε ποιο είναι ο κατάλληλος τρόπος για να υλοποιηθούν όλα αυτά τα πράγματα. Ο συνάδελφος κ. Κόχ αναφέρθηκε σε αυτά τα ζητήματα είμαι και μέλος της Επιτροπής των Μεταφορών και θα ήθελα να του ζητήσω να διερευνήσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μεταξύ των δύο επιτροπών. Χρειαζόμαστε συνέργειες. Η συνέργεια είναι ζωτική σημασία για τη δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και έτσι βλέπω ότι θα πρέπει να πορευτούμε στο μέλλον. Καλώς. Θα έχουμε λοιπόν αυτή τη συνεδρίαση, μετά οι συντονιστές θα ε, συνεδριάσουν και ο κύριος Κόχ και οι υπόλοιποι θα πρέπει να εκφράσουν ε, την μεγάλη μας επιθυμία να συνεργαστούμε με την Επιτροπή για τις Μεταφορές για αυτό τον πολύ σημαντικό φάκελο. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν για αυτά. Σήμερα θα ψηφίσουμε λοιπόν για την ε, εταιρική διακυβέρνηση. Η κυρία Λεγκρίπ καθυστέρησε, δυστυχώς. Λόγω των καλωδίων χαλκού που κλάπηκαν στο ταλής, όπως γνωρίζετε, <coughs> Όμως, ε, μου είπε η κυρία Λεγκρυπ ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με την ε, ψηφοφορία, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά εάν χρειαστεί για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, έκθεση Λεγκρυπ Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ε, υπέρ Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 5. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Τριάντα ψήφισαν. 38 τώρα. Αλλά μόνο 36 έχετε ψηφίσει. 37 ψήφισαν. Απορρίπτεται. 22 υπέρ, 16 κατά. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία παριθμών 2 υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 11, de Jong. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, άρχεται ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 11. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Σμιτ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. εγκρίνεται. 19 υπέρ, 18 κατά. Άρα οι τροπολογίες 14 και 15 καταπίπτουν. Πάμε στην 16. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 17. Τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 18. Άρχεται η ψηφοφορία. 39 μέλη. Είναι παρόντα. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται 25 προς 11. Τροπολογία 20. De Jong. Άρχεται η ψηφοφορία. ή να, από τους σοσιαλιστές κάποιος να βγάλει την κάρτα του, γιατί έχετε βάλει μία παραπάνω πριν ε, κλείσω την ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21, De Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 22, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρα 23, 24 και 25 τροπολογίες καταπίπτουν, 29 επίσης. Τροπολογία 26 Σμιτ, κατά τμήματα. Μας έχετε στείλει τον κατάλογο ψηφοφοριών, δεν θα το διαβάσω. Πρώτο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο μέρος της τροπολογίας αυτής, 26. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τρίτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 27. Τροπολογία. De Jong. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 28. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 30. Γιόγκ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 31. Τροπολογία 31 De Jong. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Για μία ψήφο. 19 προς 18. Τροπολογία 34 κατά τμήματα της, κυρία Βάιλ, της κυρίας Βάιλ. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Πέρας. 19 υπέρ, 19 κατά, άρα πίπτη. Τροπολογία 32. Κυρία Μακλάκιν. Έναρξη ψηφοφορίας για το πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται σαφέστατα. Η τροπολογία 33 καταπίπτει και πάμε στη 35. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ένας δεν ψηφίζει. Πέρα στη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 37 υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Ευχαριστούμε την κυρία Λεγκρίπ, την απουσία της. Σας ευχαριστώ όλους. Πριν μας αφήσετε να σας πω ότι θα έχουμε πολύ σημαντικά ε, project στο μέλλον. Να καλωσορίσω δύο νέα μέλη της, Ευρωπαϊ... της Επιτροπής μας μάλλον, τα οποία βλέπω εδώ τον κύριο Χατζημαρκάκη. Είναι νέο μέλος της Επιτροπής μας. Καλωσορίσατε κύριε Χατζημαρκάκη. Και τον ε, κύριο Κοφεράτη ο οποίο είναι και εκείνο καινούριο μέλο στην Επιτροπή μας. Καλώς ήλθατε κύριε Κοφεράτε. Είστε και οι δύο ευπρόσδεκτοι, ελπίζουμε να συμβάλλετε τα μάλα στις εργασίες μας. Προχωρούμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Να ξεκινήσει μια διαδικασία για τη δική μου έκθεση για τα σκάφη αναψυχή και τα ατομικά σκάφη. Επομένω, όποιος δεν έχει σχέση με το αντικείμενο, παρακαλώ να εξέλθει τις αιθούσεις και να εξέλθει σύγχος τη αιθούση. γιατί πρέπει να προχωρήσουμε και να ακούσουμε τις παρουσιάσεις για την αξιολόγηση του αντικτύπου. Λοιπόν, παρακαλώ. Uh, this is... Uh, Πρόκειται για μια σημαντική αναθεώρηση μιας οδηγίας της εσωτερικής αγοράς. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι εδώ ο συγητής από την Επιτροπή Μεταφορών, ο κύριο, κύριος Ρόμπερτ Ζήλα και ο εισηγητής Επιτροπής Περιβάλλοντος, ο κύριος Ταρταρέλα. Χαίρομαι που βρίσκονται εδώ και ελπίζω να λάβουν μέρος και στη συζήτηση ε, ταξιολόγησης επιπτώσεων ο κύριος Φαμπ, ο κύριος Ρέκο, ο κύριος Μάντερς, ο κύριος Ρούλετς είναι, είναι και ο κύριος Ντεγιόν που ελπίζω να επιστρέψει στην αίθουσα είναι οι σκιώδεις εισηγητές. Χαιρετίζω επίσης και τον κύριο Τσιράου από τη Γενική Διεύθυνση Enterprise από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι υπεύθυνο για την πρόταση αυτή θα μας πει μερικά πράγματα για το χρονοδιάγραμμα. Όπως ξέρετε με σοβαρά θέματα σαν κι αυτά ε, ξεκινούμε πρώτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρουσιάσει την αξιολόγηση αντικτύπου που έχει κάνει και οπότε ε, δίνω το λόγο τώρα στην Κομισιόν, θα κάνετε μια ε, παρουσίαση φαντάζομαι και από εκεί και πέρα θα πάρω εγώ ως εισηγητής το λόγο όπως και οι σκιώδεις εισηγητές. Ο κύριος Τζιράου λοιπόν της Κομισιόν έχει το λόγο. <coughs> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να παράσχω κάποιες εξηγήσεις όσον αφορά τις, αλλαγές ε, της οδηγίας που είναι υποσυζήτηση μετά από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την νομοθεσία που διέπει την οδηγία για τα σκάφη αναψυχής. Ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις διαφάνειες κιόλας. Βέβαια, με τον διαθέσιμο χρόνο θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σύντομοι κάνοντας μια συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης και της ανάλυσης ε, ε, ε, αντίκτυπου και με όλη την ανάλυση η οποία ε, είναι υποσυζήτηση. Κατά βάση λοιπόν θα εστιάζουμε σε τρία σημεία. Κάποιες γενικέ προφορίες ό,τι αφορά τον τομέα, ποια είναι η νομοθεσία που διέπει τον τομέα και ποιες είναι οι αλλαγές οι οποίες προτείνονται. Σε σχέση με τον τομέα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε κάποια στατιστικά στοιχεία. Η οδηγία αυτή αφορά σε 270.000 άτομα τα οποία απασχολούνται στον ε, τομέα αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνολικές ε, πωλήσει ε, είναι αξίας 9,2 δις ευρώ. Έχουμε 2.600 ναυπηγούς σκαφών ε, αναψυχής και 400 κατασκευαστές ε, μηχανών για τα σκάφη αυτά. Είναι επίσης ένας τομέας ο οποίος έχει πάρα πολύ σχηρά εξαγωγικό χαρακτήρα με διατλαντικές, με το ισοζύγιο προμόνο αν θέλετε, να είναι της ε, τάξης, ο λόγος αυτός, 3 προς 1. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι επλήγει πάρα πολύ σχηρά ο τομέας αυτός από την οικονομική κρίση του 2008-2009 με όπου πλέον οι, οι πωλήσει ε, στην πράξη σταμάτησαν. Κάποια σχετική ανάκαμψη υπήρξε το 2010 και το 2011, αλλά πόρο απέχουμε από τα επίπεδα παραγωγής που είχαμε πριν την, ε, την κρίση, πρωτού επέλθει κρίση. Σε σχέση λοιπόν με την τρέχουσα νομοθεσία. Ο στόχος είναι να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στην οδηγία 94-25 της Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στόχος λοιπόν ήταν να δημιουργηθεί μια εσωτερική αγορά για τα σκάφη αναψυχής και να εναρμονιστούν οι απαιτήσει ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Το εύρος της οδηγίας καλύπτει και τα σκάφη αναψυχής, τα ατομικά σκάφη, τα εν μέρη ολοκληρωμένα σκάφη, τις ε, μηχανές προώθησης, και μια σειρά ε, ανταλλακτικών που περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένη κατάλογο. Εξαιρεί από το ε, πεδίο της τα κανό, τα καγιάκ και τις ε, σανίδες σερφ τα ιστορικά σκάφη, τα, σκάφη, τα αγωνιστικά σκάφη και τα πειραματικά σκάφη και άλλα τα οποία κατασκευάζονται για καθαρά προσωπική χρήση και δεν τοποθετούνται, δεν μπαίνουν ποτέ για αγοραπολισία στην αγορά. Η νομοθεσία αυτή είναι μια οδηγία νέας προσέγγισης, το οποίο σημαίνει δηλαδή ότι θέτει τις βασικές προδιαγραφές και προδια... βασικές απαιτήσει μέσω των οποίων καθορίζονται τεχνικές λεπτομέρειες μέσω εναρμονισμένων προτύπων. 60 ουσιαστικά πρότυπα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 60 ε, πρότυπα τα οποία είναι ήδη σε εφαρμογή. Σε σχέση με τις ε, απαιτήσει σε σχέση που πρέπει να, να μελετηθούν, να ληφθούν υπόψη για την συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των σκαφών αυτών, πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε μία από τις τέσσερις κατηγορίες που, που δίνεται ε, ε, αφορούν στην ε, δύναμη του ανέμου και το ύψος των ε, κυμάτων. Πρέπει να ληφθούν λοιπόν αυτές οι προδιαγραφές όταν σκέφτονται τις βασικές προδιαγραφές, αυτές οι, συνθήκες όταν σκέφτονται τις βαθικές ε, απαιτήσει. Σε σχέση με την οδηγία του, υπάρξαν μια καταρχήν μεταρρύθμιση το 2003 όπου διευρύνθη το εύρος της αρχικής οδηγίας του 1994 για να συμπεριλάβει τα ατομικά σκάφη και τις μηχανές προώθησης. Ε, επίσης εισήγαγε ε, τη λεγόμενη ε, αξιολόγηση συμμόρφωσης μετά την καταστροφή, ώστε, μετά την, κατα, μετά την κατασκευή, ώστε να λαμβάνει υπόψη και εισαγόμενα σκάφη και εισαγόμενα ανταλλακτικά από, τις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για καταναλωτές οι οποίοι για παράδειγμα ανήκουν σε ιστιοπλοϊκούς ομίλους κλπ. Αλλά που δεν ε, ε, αποκτούν τα σκάφη τους μέσω του συνήθους εμπορικού κυκλώματος και ήταν σημαντικό να συμπεριληφθούν και αυτά τα σκάφη στο εύρος της ε, οδηγίας. Και η τροπολογία αυτή του 2003 επίσης σήγαγε και περιβαλλοντικές συνθήκες σε ό,τι αφορά τις εκπομπές, τις, τις ρηπαίνουσες εκπομπές των μηχανών και τις και την ε, εκπομπές θορύβου. Και επίσης έλαβε, ε, έλαβε υπόψη και νέες τεχνικές προδιαγραφές. Ποιε είναι λοιπόν οι βασικές ε, απαιτήσεις. Υπάρχουν οι γενικές, οι οποίες δίνουν διάφορες διαγραφές σε ό,τι αφορά την, την εμφάνιση της την εμφάνιση των πινακίδων της, ε, του ναυπηγού, την ε, ε, αναγνώριση του κήτους, την σχετική, το, σχετικό, το σχετικό εγχειρίδιο ιδιοκτήτη κλπ. Και επίσης να συμπεριλάβει διάφορες, διάφορα θέματα που αφορούν στην, στις κατασκευαστικές προδιαγραφές. έτσι, η έκθεση αξιολόγησης συμμόρφωσης προς τις ε, προδιαγραφές, ε, διαφοροποιεί τις απαιτήσει που υπάρχουν για τα σκάφη με μήκος λιγότερο των 12 μέτρων και μεγαλύτερο από αυτά, αλλά πάντως ε, υπάρχει ουσιαστικά και μια δυνατότητα αυτοτελούς προσωπικής υποβολής έκθεσης σε ό,τι αφορά την συμμόρφωση. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει η παρέμβαση της ε, έκθεσης ε, αξιολόγησης των τροποποιήσεων που μπορεί να έχουν επέλθει σε ένα σκάφος και που αξιολογεί το σε διάφορες προδιαγραφές και το τι έχει συμβεί σε ό,τι αφορά τα στατικά μέρη και τα ανταλλακτικά. Υπάρχει δυνατότητα για προσωπικά σκάφη, επίσης ε, ατομικής η διαβουλήση δήλωση σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση και υπάρχουν βέβαια πιστοποιημένα όργανα τα οποία παρεμβαίνουν για να, κάνουν τις σχετικές, να συντάξουν τις σχετικές εκθέσεις ε, συμμόρφωσης. Και σε ό,τι αφορά τις εκπομπές ε, θορύβων, την ηχορύπανση δηλαδή, αξιολογείται η συμμόρφωση αλλά και στο παρελθόν, αλλά οι περισσότερες βέβαια αυτού του είδους εκθέσεις απαιτούν την παρέμβαση πιστοποιημένων οργάνων. Τώρα, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή για την προετοιμασία της μεταρρύθμισης τους νόλους οδηγίας αυτής. Η όλη, η όλη προετοιμασία ξεκινήσε το 2004 με μια άσκηση απογραφής, με την πρώτη μελέτη ε, ε, ε, αξιολόγησης του αντίκτυπου το 2006, με μια έκθεση της Επιτροπής του 2007, μια συμπληρωματική έκθεση αξιολόγησης του αντίκτυπου το 2008 και με δημόσια διαβούλευση, η οποία ξεκίνησε το 2009 και μέρος του 2010. Οι κυρίες αλλαγές λοιπόν ποιες είναι. Κατά βάση, δύο προσεγγίσεις ελάφθησαν υπόψη. Η μία να αξιολογηθεί τι, ποιες θα μπορούσαν να είναι οι αλλαγές ή τι απαιτείται σε σχέση με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας αυτής και το άλλο είναι το ποιες μπορεί να είναι οι αλλαγές που είναι απαιτούμενες σε σχέση την ε, το κομμάτι το περιβαλλοντικό και τη συγχωρήπανσης σε ό,τι αφορά την οδηγία. Σε σχέση βέβαια με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην νομοθεσία, έτσι λοιπόν μια πρώτη αξιολόγηση που έγινε ουσιαστικά αναγνώρισε ότι πρέπει υπάρχει ανάγκη διευκρίνησης κάποιων ορισμών σε ό,τι αφορά το εύρος της ε, ε, οδηγίας. Πρέπει να υπάρχει μια διευκρίνηση σε ό,τι αφορά την, μετά την κατασκευή αξιολόγηση και σε ποια σκάφη θα πρέπει να εφαρμόζεται. Υπήρξε, εντοπίστηκε επίσης η ανάγκη ευθυγράμμισης της οδηγίας στο νέο ε, νομικό πλαίσιο και επίσης η νέα αυτή οδηγία να συνάδει προς την ε, ε, σύμβαση σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά στοιχεία και την ανομοθεσία που έχει εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στη συνέχεια αναγνωρίστηκε η ανάγκη μεταρρύθμισης και βελτίωσης των περιβαλλοντικών ε, επιδόσεων των σκαφών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις δυνατότητες να προαχθεί η ανταγωνιστικότητα αυτού του τομέα. Σε σχέση λοιπόν με το εύρος εφαρμογής, με το πεδίο εφαρμογής, με το πεδίο εφαρμογής της ε, νέας οδηγίας, θέλω να επαναλάβω ότι δεν υπάρχουν μίσονες αλλαγές σε ό,τι αφορά το σημείο αυτό. Οι νέες διατάξεις είναι κατακλείδη διευκρινιστικές διατάξεις. Είναι μόνο τα ατομικά σκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται για να αναψυχή ή αθλητισμό και συμπεριλαμβάνονται στην ε, νέα οδηγία. Τα αμφίβια σκάφη εξαιρούνται και δεν διευκρινίζεται ότι τα κανό και τα καγιάκ που έχουν σχεδιαστεί να την χάν ε, εξαιρούνται εκτός από αυτά τα οποία προωθούνται. Εάν μόνο, συγγνώμη, εξαιρούνται εάν έχουν ως μόνο προωθητική δύναμη τον, ε, την ποδηλασία. Θαλάσσια ποδηλασία. Οι νέοι ορισμοί συγκεκριμένοι για τον τομέα αυτό που εισάγονται τώρα είναι τα σκάφη τα οποία ναυπηγούνται για ίδια χρήση, θα πρέπει να διευκρινιστούν σε σχέση με την χρήση εν μέρη κατασκευασμένων ε, κομματιών του σκάφους και μια άλλη σε ένας άλλος σημαντικός ορισμός ε, αφορούσε σε ιδιώτες εισαγωγής και συνδέεται η, διάταξη αυτή με την αξιολόγηση του σκάφους και των επιδόσεών του μετά την κατασκευή. Και όλα αυτά βέβαια αυτά συνδέονται με το κατά πόσον ε, όλα αυτά συνδέονται με καθαρά ατομική χρήση. Σε σχέση λοιπόν με την ευθυγράμμιση της οδηγίας στο νέο νομικό πλαίσιο, υπάρχουν πλέον δύο ε, οριζόντιοι ε, κανόνες που είναι πασίγνωστοι, ε, δύο νομικά πλαίσια. Ο κανονισμός 765 κάθετος 2008 και η απόφαση του Συμβουλίου της 9 η Ιουλίου του 2008 που αφορούν στις απαιτήσει για την πιστοποίηση και εποπτεία της αγοράς σε σχέση με την εμπορία των προϊόντων αυτών Στη συνέχεια, σε σχέση με τα όρια εκπομπών, ελήφθη υπόψη η ανάγκη για πολύ πιο αυστηρά καθορισμένα όρια σε ό,τι αφορά τις εκπομπές, αλλά πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας την συνεισφορά των σκαφών αναψυχής στην ηχορύπανση σε σχέση με τις συνολικές εκπομπές που είναι, σχεδόν, που είναι 0,20% ενώ οι συνολικές εκπομπές είναι 0,1%. Τα σενάρια λοιπόν τα οποία θα εξετάσουμε σε σχέση με, τις, ε, με, τις, ε, με τα πρότυπα για τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές θα αφορά μόνο την εκπομπή οξυδίων του αζότου εάν ξεπερνούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα εκπομπών σε σενάριο πολύ υψηλών συγκεντρώσεων ασκαφών ψυχής στην ίδια ζώνη, στα ίδια λιμάνια και τις ε, στιγμές ακριβώς τις ώρες ε, κορύφωσης του φόρτου. Λαμβάνει επίσης υπόψη πολύ πιο αυστηρά πρότυπα σε ό,τι αφορά άλλες περιοχές ώστε να εξετάσουμε τι μπορεί να... άλλα πεδία για να δούμε τι μπορεί να προταθεί στα πλαίσια αυτής της αναθεώρησης. Τρία σενάρια λοιπόν αξιολογήθηκαν. Η πρώτη εναλλακτική ήταν να συνεχίσουμε όσα έχουμε και να μην υπάρξει καμία αλλαγή. Ένα δεύτερο σενάριο που θα έλαβε υπόψη την εισαγωγή πολύ πιο αυστηρών ορίων ε, ε, ρηπαντικών εκπομπών και το τρίτο σενάριο εξετάζει πολύ πιο αυστηρά όρια ε, ρηπογόνων εκπομπών συνδυασμένων με μέτρα απάλυνσης του φαινομένου. Με τρεις ε, υποενότητες το σενάριο αυτό. Το πρώτο τη χρήση ενός σχεδίου ευελιξίας, το δεύτερο την εισαγωγή μιας περίοδου ε, ε, μεταβατικής περίοδου για όλους και η τρίτη εναλλακτική τη χρήση μιας μεταβατικής περίοδου για όλους τους ναυπηγούς, για όλους τους κατασκευαστές ε, μηχανών, αλλά και πιο συγκεκριμένη μεταβατική περίοδο για τους ε, μικρομεσαίους ε, ναυπηγούς. Σε σχέση λοιπόν με την αξιολόγηση της κατάστασης έχει και την ε, μελετώμενη μεταρρύθμιση, το δεύτερο σενάριο, σε σχέση δηλαδή με την εισαγωγή πολύ πιο, μόνο πολύ πιο αυστηρών ορίων ε, ρηπαντικών ε, εκπομπών, ε, προβλέπει ένα καθαρό όφελος 1,9 έως 34,1 εκατομμυρίων ευρώ, με το πολύ πιο αυστηρό σενάριο, στο, στην πρώτη υπολύση, ε, το, το πρώτο υποσενάριο ε, δίνει ένα καθαρό όφελος 4,8 με 34,6 εκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο υποσενάριο με την χρήση μιας μεταβατικής περίοδου αυξάνει τα ωφέλη αυτά, ώστε να έχουμε ένα καθαρό κέρδος 5,7 έως 34,9 εκατομμυρίων ευρώ. Και το τρίτο υποσενάριο με τη χρήση μεταβατικής περίοδου, δηλαδή που επεκτείνεται σε όλες τις μικρομεσαίες ε, ναυπηγικές ε, ε, επιχειρήσεις και τις κατασκευαστές εξολέμβιων μηχανών. Το κέρδος είναι 5,7 με 34,8 εκατομμύρια ευρώ. Σε σχέση τώρα με τον κοινωνικό αντίκτυπο, ε, ανάλογα με την υιοθέτηση οποιασδήποτε από τις προηγούμενες λύσεις. Υπάρχει πάντα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των ε, εξολέμβιων μηχανών σε ένα e CD2. Έχουμε για αυτές τις περιπτώσεις ε, απώλειες θέσεων εργασίας με το δεύτερο υποσενάριο, γιατί στο πρώτο δεν έχουμε καμία αντίκτυπο σχετικό, ε, απώλεια λιγότερων από 100 θέσεις απασχόλησης για την ε, υπολύση 3,2, δηλαδή με, το, μεταβατική περίοδο, είναι πολύ απίθανη απώλεια θέσεων απασχόλησης και για τις ε, μηχανές SI λιγότερες από 100 οι θέσεις απασχόλησης που χάνονται και για το πολύ αυστηρό σχέδιο, το τρίτο υποσενάριο, με το πιο αυστηρά κριτήρια που εισάγονται αλλά και μεταβατική περίοδο, είναι απίθανο να χαθούν θέσεις απασχόλησης είτε για τον πρώτη, είτε για την περίπτωση CI, είτε για την περίπτωση SI μηχανών. Και όταν παρατείνουμε την μεταβατική περίοδο για τις μικρομεσαίες ναυπηγικές ε, ε, επιχειρήσεις και στις δύο περιπτώσεις είναι απίθανη η απώλεια θέσεων απασχόλησης. Το συμπέρασμα λοιπόν, τα συμπεράσματα μάλλον είναι τα ακόλουθα. Συγγνώμη, λέει ο όχι. Αξιολογήθηκε επίσης η τρέχουσα κατάσταση και η πιθανότητα μείωσης των, της συγχωρήπασης. Σε σχέση με την χορύπανση υπάρχει ανάγκη να ληφθεί υπόψη ότι η χορύπανση από τα σκάφη αναψυχής δεν συνδέεται μόνο με τις μηχανές, έτσι αρθρώνονται λοιπόν από ένα συνδυασμό παραγόντων, όπως τον τύπο του κήτους του σκάφους και τις ε, φυσικές συνθήκες, όπως είναι η ένταση του ανέμου, τα, το μέγεθος των κυμάτων κλπ. Και πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι η αντίληψη ε, θορύβου δεν είναι αντικειμενικό στοιχείο, είναι υποκειμενικό σε ό,τι αφορά την αντίληψη αυτής της χορύπωνσης, που εξαρτάται πολύ κατά πόσο βρισκόμαστε σε πρωινές ή νυχτερινές ώρες, σε σχέση με την τοπογραφία του, του τόπου κλπ. Η μείωση λοιπόν της συγχωρήπανσης για ό,τι αφορά τις μηχανές των σκαφών αναψυχής, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι καταχάς συνεισφέρει μόνο σε πολύ μικρό ποσοστό στον ε, ε, θόρυβο που γίνεται αντιληπτός και το όφελος από την περαιτέρω μείωση των ορίων ηχορύπανσης που προβλέπονται αυτή τη στιγμή από την αποθεσία είναι πάρα πάρα πολύ ε, μικρός, πάρα πολύ χαμηλός σε σχέση με τα κόστη τα οποία θα συνεπαγόταν ο επανασχεδιασμός της εξολέμβιας μηχανής προκειμένου να υπάρξει από τον κινητήρα και μόνο από τη μηχανή μείωση του θορύβου λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα υπάρξει αναλογικό όφελος σε ό,τι αφορά τον ανταλαμβανόμενο κίνδυνο, τον αναλαμβανόμενο συγγνώμη, τον, την ανταλαμβανόμενη ηχορύπανση από τους καταναλωτές. Εξετάσαμε ποιες, είναι, ποιες άλλες είναι οι διατηθέμενες ε, εναλλακτικές για να μειωθεί η χορήμανση των, των, ε, των ατομικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής. Οι, οι πιθανότητες συνδέονται εν με την μείωση ταχύτητας σε κάποιες περιοχές και το, και το άρθρο 4 σημείο 5 της προτινόμενης οδηγίας ε, προβλέπει σε συγκεκριμένες περιοχές την υιοθέτηση αυτού του ορίου η χωρικανσίες που θα επιτρέπει επομένως να υπάρξει μία μείωση του θορύβου που χρησιμοποιεί τη χρήση των εργαλείων αυτών. Η εναλλακτική στη συνέχεια ήταν σε σχέση με την μείωση των εκπομπών να χρησιμοποιηθεί η μεταβατική περίοδος για τα μικρομεσαία σκάφη σε σχέση με, τον, με τους κατασκευαστές ναυπηγούς και τους κατασκευαστές μηχανών και να μην προταθούν αλλαγές σε σχέση με τα όρια ηχορύπανσης. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτά τα όρια εκπομπών θα έχουν θετικό αντίκτυπο αυτό που περιλαμβάνεται λοιπόν στη νέα πρόταση έχει και θετικό αντίκτυπο σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα και τις θέσεις απασχόλησης. Γιατί ένα από τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία ήταν να ληφθεί υπόψη ότι υπήρχαν πάρα πολλές διαφορετικές ε, απαιτήσει ε, στην ε, επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο συνεπάγεται διαφορετικές γραμμές παραγωγής με ποικίλο κόστος για να μπορέσει να υπάρχει συμμόρφωση με τις διαφορετικές ε, προδιαγραφές και απαιτήσεις σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Αυτό που τώρα προτείνεται είναι πολύ παρεμφερές με αυτό που ισχύει σε διάφορα άλλα μέρη του πλανήτη και επομένως θα δώσετε δυνατότητα στην βιομηχανία μας να υποφεληθεί ε, οικονομιών κλίμακας και επίσης προαγωγής και καλύτερης εμπορίας των σκαφών που να φυγούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βελτιώνοντας την γενική ανταγωνιστικότητα του χώρου. Θα ήθελα να ολοκληρώσω εδώ την παρουσίαση αυτή. Σας ευχαριστώ θερμά για την, παρουσία, για την προσοχή σας και βέβαια στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση θα θέλατε να έχετε και οποιοδήποτε ερώτημα θέλατε να υποβάλλετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος για την παρουσίαση αυτή που ήδη μας βάζει μέσα στο κλίμα. Θα ήθελα να χαιρετήσω εδώ εκ μέρους της Επιτροπής μια ομάδα σπουδαστών από το Πανεπιστήμιο Άστον. Βλέπω τον καθηγητικό ψησική εκεί στο τέλος. Είναι τελ, τελείως σύμπτωση αγαπητοί συνάδελφοι το ότι έφτασα την ώρα που θα κάνω εγώ την ομιλία μου αλλά τέλος πάντων τους καλωσορίζω και χαίρομαι που βρίσκονται εδώ λοιπόν ακούσαμε το την Επιτροπή θα ακούσουμε και τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές οι περισσότεροι είναι εδώ κύριος Γιόγκ δεν είναι εδώ, δυστυχώς, αλλά τέλος πάντων, εγώ ως εισηγητής σας αρχίσω τη συζήτηση. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο που ακούσαμε αυτά που ακούσαμε για τον αξιολόγηση αντικτύπου ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με το θέμα αυτό εδώ και κάμποσο καιρό. Αναφερθήκατε επίσης στις προσπάθειες αναθεώρησης της οδηγίας που έγιναν ήδη από το 2007 έχουν ξεκινήσει και μας είπατε ακριβώς ε, θα, ήταν οι επιπτώσεις οι ναυπηγικές ε, κατασκευαστικές εταιρείε βεβαίως και οι πολίτες της Ευρώπης ε, εγώ εκείνο που θα ήθελα να πω για τα νέα όρια εκπομπής καυσίμων, εκπομπών καυσίμων είναι το εξής. Οι νέες προτάσεις για αυτά τα όρια, για τα σκάφη ε, αναψυχής ιδιαίτερα ε, αυτά συγκεκριμένα με τη εξολέ, με, που κινούνται με μηχανή ε, τα όρια αυτά λοιπόν μοιάζουν, είναι πολύ κοντά σε αυτά που εφαρμόζονται στις Ηνωμένε Πολιτείες, στην Αμερική μάλλον γενικότερα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να αρχίσουμε να βλέπουμε, να συγκρίνουμε το τι κάνουμε εδώ με το τι γίνεται εκεί. Υπάρχουν επίσης Ε, ακούσαμε κάποια σύγκριση και θα πρέπει να γίνει σύγκριση αυτή με το πακέτο General Goods ε, για να δούμε μήπως χρειάζεται να ε, αλλάξουμε ορισμένα πράγματα. Βεβαίως στον κλάδο για τον οποίο μιλάμε κατασκευάζονται πάρα πολλά σκάφη βάσει των επιθυμιών του αγοραστή. Είναι δηλαδή τελείω ειδικέ και μοναδικές κατασκευές. Δεν ξέρω αν εδώ πρέπει να γίνουν αλλαγές ή εν πάση περιπτώσει αν παραμελήθηκε το κομμάτι αυτό, το μέρος αυτό του κλάδου συνειδητά ή όχι από τα κράτη-μέλη. Ε, Αυτά από πλευρά μου. Θα δώσω το λόγο τώρα στους σκιώδεις για να κάνουν κάποια σχόλια. Α, να πω επίσης ότι οι σκιώδεις να πω ότι πρέπει να συνεργαστούμε πολύ στενά με τους σκιώδεις συγητές για να προχωρήσουμε την υπόθεση αυτή και όπως ξέρουν οι περισσότεροι από εσά θα γίνει μια διερευνητική αποστολή τρόπων για να έρθουμε σε επαφή με τους ε, κατασκευαστές ε, στο Düsseldorf την πέμπτη αυτή μεθαύριο ε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από εδώ στις 7 η ώρα το πρωί για να είμαστε και στην ώρα μας. Ελπίζω όμως να συμμετάσχετε στην αποστολή αυτή, τη διαρευνητική όπως είπα. Λοιπόν, θέλετε και εσείς να μιλήσετε βεβαίω. Ας αρχίσουμε με τους σκιώδεις συζητητές της Επιτροπής εδώ μετά κύριο Σταρδαρένα, μετά κύριο κύριος Κομφεράτη και όποιος άλλος θα ήθελε να μιλήσει ο κύριος Φαμπ ευχαριστώ πρόεδρε σας ευχαριστώ πρώτα πρώτα εσάς για αυτά που μας είπατε θα ήθελα και εγώ να πω από πλευράς μου ότι το χρόνο διάγραμμα που προτείνεται είναι καλό, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που προτείνεται και δεν υπάρχει πρόβλημα να μην γίνει τελική ψηφορία στις 8 Μαΐου. Ε, σήμερα παρόλο που ε, Τέλο πάντων χρησιμοποιώ και εγώ τα σκάφη αυτά. Προσπαθώ, θα προσπαθήσω να είμαι ουδέτερος παρατηρητής του κλάδου αυτού, του τομέα αυτού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την παρουσίαση που έκανε σήμερα το πρωί. Πρόκειται για πολύπλοκο θέμα. Ε, θα ήθελα να πω επίση ότι χαιρετίζω την εκδήλωση, την συνάντηση στο Ντιουσελντόρφ στην οποία όμως δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ διότι θα συναντήσω τους δικούς μας ε, ε κατασκευαστές ε, σκαφών στο Μπόντενζε. Αυτά που μας είπε η Κομισιόν ε, είναι σωστά, είναι αλήθεια ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις από την αναθεώρηση της οδηγίας στα οικονομικά κυρίως των κατασκευαστικών επιχειρήσεων και αυτό είναι πολύ σημαντικό ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσης. Καταλαβαίνουμε αυτό που είπατε εσείς για την Αμερική, ξέρουμε πολύ καλά που γίνονται στην Αμερική και αυτά που έκανε η Καλιφόρνια πριν από δύο χρόνια αλλά ε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και την κρίση την οποία διέρχεται η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ε, θυμάμαι από παλιότερα ε, όταν ασχολήθηκα με τα ελαστικά των ε, οχημάτων πόσο δύσκολο ήταν να υπολογίσουμε την χορύπανση. Η Κομισιόν εδώ προτείνει να μην γίνει αλλαγή το καταλαβαίνω αυτό γιατί είναι πολύ δύσκολο το θέμα. Α, θα χαιρόμαστε λοιπόν που δεν προτείνονται αλλαγέ οι οποίε θα δημιουργήσουν αταραχέ στον κλάδο. Και τρίτον, α, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα το θα ήθελα να πω για να μην καταντήξουμε να έχουμε και εμείς σκάνδαλα σαν και αυτά που έχουμε με τα εμφυτεύματα στήθους πρόσφατα στην Ευρώπη ναι, θα πρέπει, ότι θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και θα πρέπει να ελέγξουμε τη συμμόρφωση αυτής της τροποποιημένης πλέον αναθεωρημένης οδηγίας με τις άλλες συναφείς οδηγίες. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι ότι τουλάχιστον στη χώρα μου, στη Γερμανία, υπάρχουν και ιδιώτες οι οποίοι κατασκευάζουν ε, σκάφη. Ε, αθλητικά και άλλα. Ε, εδώ δεν περιλαμβάνονται αυτοί, περιοριζόμαστε στους εμπορικούς, στους εμπόρους κατασκευαστές, κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Ίσως θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη και τους ιδιώτες κατασκευαστές, αλλά σε γενικές γραμμές υποστηρίζω αυτά που ελέγχθησαν και που είπε η Κομισιόν. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι με ενδιαφέρουν βεβαίως τα σκάφη και μου αρέσει πάρα πολύ η αστιοπλοεία και νιώθω μεγάλη περηφάνεια όταν κάνω αστιοπλοεία και μπορώ να βγω από το λιμάνι χωρίς να βασιστώ στο κινητήρα και μπορώ και να επιστρέψω στο λιμάνι χωρίς κινητήρα. Για μένα αυτό είναι το καλύτερο. Από την άλλη δεν μπορούμε να αμελήσουμε ε, τους κινητήρες, τις εξολέμβιες μηχανές Εξού και είναι πολύ σημαντικά ε, τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος στα οποία θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα. Όταν μιλούμε για σκάφη αναψυχής, θα πρέπει να πούμε ότι όταν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα, έχει επιπτώσεις που κρατούν πολύ σε βάθος χρόνου και γι' αυτό θα πρέπει να είναι πιο αυστηρά τα όρια εκπομπεών των ρήπων για να βελτιωθεί η ποιότητα των υδάτων, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να βελτιωθεί και η ανταγωνιστική μας θέση γενικότερα. Ως προς την ηχορύπανση, από πείρας μπορώ να σας πω ότι οι εξολέμβιες μηχανές που θα ενσωματωθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αφορούν κυρίως τα διάφορα jet ski τα οποία ε, πλέουν πάρα πολύ κοντά στις ακτές και κάνουν πάρα πολύ θόρυβο. Και γι' αυτό εγώ έχω συναντηθεί με φορείς της ιδιωτικής αγοράς που εκπροσωπούν τον ε, κλάδο αυτό ε, και χαίρομαι πάρα πολύ διότι έχει ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος και στις θέσεις απασχόλησης αλλά και ο αντίκτυπος στην κοινωνία γενικότερα. Είμαι πεπισμένος ότι υπό την ε, διεύθυνση του Προέδρου κυρίου Μάλκολμ Χάρμπορ θα καταφέρουμε να διαδραματίσουμε πολύ σημαντικό ρόλο και θα καταφέρουμε να ενισχύσουμε την αηφόρο ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you very uh, Κύριος Μάντερς, ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εισαγωγή που έκανε. Η πρόταση είναι ξερά ισορροπ... αρκετά ισορροπημένη. Βεβαίω, ε, συμφωνώ με αυτό που είπατε και εσεί, Θα πρέπει να δούμε ε, παγκοσμίως τι γίνεται. Ε, ιδιαίτερα τώρα που υπάρχει ε, κρίση. Γιατί είναι σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε εξαγωγέ από την Ευρώπη. Και Πραγματικά πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμπλέκονται εδώ, άρα αν είχαμε ε, κανόνες παγκόσμιους ε, που να ίσχυαν παντού θα βοηθούσαμε τις εξαγωγές. Τώρα για τα σκούτερ αυτά ή τα jet ski που αναφέρατε, Όντως αυτά τα ατομικά σκάφη είναι τα πιο προβληματικά όσον αφορά το θόρυβο την ηχορύπανση. Εδώ τώρα μιλάμε για θέση σε εμπορία, θε, κυκλοφορία στην αγορά. Εκείνο που είναι σημαντικό ή ε, όμως Νομίζω ότι δεν είναι να αναφέρουμε αυτό γιατί είναι πιο εύκολο ένας ιδιώτης να το πάρει το σκάφος αυτό και να το εισάγει από μόνος του. Εκείνο που, για το οποίο θα πρέπει να μιλάμε είναι η χρήση στην Ευρώπη. Τώρα, βενζίνα ή ντίζελ σε ορισμένες χώρες ε, επιτρέπεται η διζελ σε της βενζίνας ε, και του ντίζελ παντού και στα σκάφη ίσως θα πρέπει να το δούμε βέβαια όχι ότι εντάσσεται σε τούτη την οδηγία αλλά θα πρέπει να ε, να το δούμε κάποια στιγμή το θέμα αυτό και ξέρετε ότι για τα τρακτέρ φωνάζω να υπάρχει μία και μόνη ενιαία άδεια τώρα για τα σκάφη δεν είπαμε ότι είναι άμεσα επίγον το θέμα αλλά κάποτε πρέπει να το συζητήσουμε σίγουρα λέει ο πρόεδρος δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε τώρα ίσως να πρέπει να το δει η Επιτροπή Μεταφορών αυτό γιατί εκείνη είναι πιο αρμόδη για την ασφάλεια και τα λοιπά. Δεν ξέρω και αυτοί ασχολήθηκαν και με τους οδηγούς των σιδηροδρόμων και με τα κράνια για τους μοτοσυκλετιστές και τα λοιπά. Η κυρία Κράνεν, δεν χρειάζεται να επαναλάβω όλα αυτά που ελέγχθησαν. Ε, εκείνο το οποίο συμφωνώ με, ε, με αυτά που ελέγχθησαν και με τις ερωτήσεις του κυρίου Μάντερς δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο εκείνο το οποίο θέλω να πω μοναχά είναι νομίζω ότι όλοι μπορεί να συνεργαστούμε και με την Επιτροπή Μεταφορών θα πρέπει να συνεργαστούμε πολύ καλά και οι παρουσίες της Κομισιόν ήταν πάρα πολύ καλή τώρα ο κύριος Ζήλερ μετά ο κύριος Ταταρέλα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να παρακολουθήσω τη συζήτηση και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και την Κομισιόν για την παρουσίαση που μας ε, έκανε δεν αρχίσαμε βεβαίως ε, τη συζήτηση στην Επιτροπή Μεταφορών αλλά όπως κάναμε και παλιότερα θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην ασφάλεια γιατί αυτή είναι κύριο μέλημά μας στην Επιτροπή Μεταφορών νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να πάρουμε αποφάσεις και μέτρα τα οποία να ε, συντηρούν αν θέλετε να διατηρούν την ανταγωνιστικότητα του, των επιχειρήσεών μας. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά λόμπι ε, που πιέζουν για να ε, εντάξουμε στο πεδίο εφαρμογής ή να αποκλείσουμε από το πεδίο εφαρμογής κάποιες κατηγορίες καφών ε, θυμάμαι δεν έχουμε συζητήσει πολλά περί αυτού στην Επιτροπή Μεταφορών αλλά σίγουρα θα τα συζητήσουμε αυτά. Τώρα για τις, ε, τα όρια εκπομπών καυσίμων αφενός που επιλέγεται την εναλλακτική 3-3 και για τον χωρί λέτε να μην υπάρξει καμία αλλαγή συμφωνούμε ή μάλλον σημειώνουμε το τι ε, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το συζητήσουμε κι εμείς. Ο κύριος Ταρταρέλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν πάρα πολύ σύντομο, πάρα πολύ ε, χρήσιμο που βρέθηκα εδώ και να παρακολουθήσουμε την ε, εισήγηση αυτή που έγινε και από τον εισηγητή και από την Επιτροπή. Πρόκειται για έναν θύλακα θέλετε της αγοράς, αλλά εξαιρετικά σημαντικό και που είναι σημαντικό να τον υποστηρίξουμε και να τον βοηθήσουμε. Εμείς στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για τις πτυχές οι οποίες αφορούν το περιβάλλον η δική μου άποψη σε ό,τι αφορά την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι θετική, γιατί βρίσκομαι σε μια επιτροπή που ε, έχουμε, έχουμε βρεθεί σε αμηχανία και ε, σε σύγχυση πολλές φορές στο θέμα αυτό. Αν θέλετε, ε, βρισκόμαστε σε μια θάλασσα αρκετά ε, ταραγμένη ανάμεσα στα ζητήματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, την ανάπτυξη, αλλά από την άλλη πλευρά την αναγκαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος. Όμως, επαναλαμβάνω, κατά βάση η άποψή μου είναι θετική για την πρόταση. Με μια μεγαλύτερη προσοχή που ίσως θα επιθυμούσα να ζητήσω πάνω στο πρόβλημα της χορύπανσης. Βλέπω ότι η Επιτροπή το επιλύει το ζήτημα μόνο με μια μείωση της ταχύτητας των σκαφών. Όμως το θέμα μείωση ταχύτητας είναι ένα πρόβλημα το οποίο άπτεται της ασφάλειας και εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Αλλά μια περαιτέρω προσπάθεια πάνω στη θεματική της μείωσης της ηχορύπανσης, εγώ θα την επιθυμούσα. Γιατί ανάμεσά μας, όλοι μας, αλλά και γενικά αν θέλετε, οποιοδήποτε ασχολείται με τα ζητήματα αυτά, υπάρχει πολύ μεγάλη υποτίμηση του προβλήματος της συγχωρήπανσης και πιθανότητα δεν είναι ορατό και δεν αντιλαμβάνεται το θέμα αυτό όπως άλλοι τύπου ρήπανσης. Όμως τονίζω ότι η χωρήπανση επηρεάζει άμεσα το άτιμο και η ρήπανση του περιβάλλοντος έχει ευρύτερη ε, επιρροή και αντίκτυπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλια αυτά. Άλλο μέλος που θα ήθελα ήσταν ήδη στο κατάλογο των εισηγητών. Κύριε Πρόεδρε, η εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή η εργασία αναθεώρησης, ήταν εξαιρετικά σημαντική. Αλλά ακριβώ γι' αυτό, τόσο κατά στα μάτια μου όσο και στα μάτια άλλων συναδέλφων, φαίνεται πολύ πιο ισχυρή τα, ισχυρά τα όρια τα οποία προκύπτουν από την έλλειψη ενός, ε, δεσμε, μιας δεσμευτικής ε, ε, νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την χορύπανση. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα σκάφη αναψυχής. Είναι αδύνατο να μιλήσουμε για προστασία του περιβάλλοντος όταν μαζί με τις ρηπογόνες εκπομπής και όλων των στοιχείων που διακυβεύουν την ασφάλεια χρήση των μέσων αυτών συνδέεται και το θέμα της Πρόκειται, υπάρχουν σκάφη τα οποία ε, κυκλοφορούν, αν θέλετε, ε, κινούνται πολύ κοντά στις ακτές και που κανονικά ακόμα και τα πλέον σύγχρονα σκάφη εξακολουθούν να έχουν ένα επίπεδο ηχορύπανσης υπερβολικά υψηλό. Και πραγματικά θεωρώ ακατανόητο. Ακόμα και με τις παρατηρήσεις που έγιναν από την Επιτροπή, δεν είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχουν τεχνικά μέσα για να, για να γίνει απολογισμός και αντικειμενική εκτίμηση του επίπεδου της χορύπανσης. Στην, ε, θα έδινε πολύ μεγαλύτερη ισχύ και μεγαλύτερη δύναμη και ανταγωνιστικότητα στην ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία ναυπήγησης αν εισάγαμε και αυτούς τους όρους. Γιατί μετά από μια αρχική δύσκολη κατάσταση στη συνέχεια θα ήταν η πολύ πιο αντιγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία γιατί σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου δεν ασχολούνται με το καθορισμού καθορισμό ακριβώς αυτών των ορίων ηχορύπανσης. Θα ζητούσα λοιπόν ε, έντονα μια καλύτερη θέαση του θέματος, γιατί μια τόσο καλή δουλειά δεν μπορεί να έχει ένα κενό. Παραδόξως, όσο πιο ολοκληρωμένη είναι μια εργασία και δεσμευτική, τόσο μεγαλύτερο κενό και χάσμα βλέπουμε σε άλλα πεδία. Θα ήθελα να κάνω μόνο μία παρατήρηση και σε μια άλλη θεματική που αφορά την αυτοδήλωση, την αυτοπιστοποίηση. Από άψη διαδικασιών αυτή η αυτοπιστοποίηση είναι να αμφισβήτα ο δρόμος ο οποίος ε, απλοποιεί τα πράγματα και τα κάνει πολύ πιο γρήγορα. Αλλά πρέπει να ληφθούν, να ληφθούν απόψη κάποιον. Δηλαδή οι κυρώσεις θα πρέπει να γίνονται πάρα πάρα πολύ ε, αυστηρές. Γιατί η κύρωση η οποία καθορίζει αν θέλετε την αποθάρρυνση και επομένως την πραγματική αντιδιαστολή με μια δράση που μπορεί να είναι μορφής απλής ανακοίνωσης, καταγγελίας ανακοίνωσης πραγματικότητας. Εάν θέλουμε δηλαδή να διατηρήσουμε την πράξη αυτοπιστοποίηση, καταλαβαίνω τους λόγους, θα πρέπει σε περίπτωση καταγγελίας οι κυρώσεις να είναι πάρα πολύ αυστηρές για να υπάρχει ουσιαστική αποθάρρυνση των παραβατών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα σχόλια. Θα γίνει μια σύντομη σύνοψη στο τέλος, αλλά πάντως μπορεί το Προεδρείο να, να κάνουμε μια σύνοψη όλων των αποτελεσμάτων. Νομίζω ότι το θέμα της συγχωρήπασης είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Και βεβαίως θα καλυφθεί στο κείμενό σας. Θα σας δώσω το λόγο λοιπόν για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να επιβεβαιώσω ότι πράγματι το τμήμα της πρότασης που έχει να κάνει με το περιβάλλον είναι πολύ παρεμφερές με το υφιστάμενο πλαίσιο στις Ηνωμένε Πολιτείες. Πράγματι προσπαθούμε να διατηρήσουμε και να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα και να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε τις θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σεβόμαστε πλήρως το νέο νομικό πλαίσιο, θα πρέπει να υπάρξει ευθυγράμμιση. Έχουμε θεσπίσει την έννοια του ιδιώτη εισαγωγέα. Συζητείτε βεβαίως η έννοια αυτή Ωστόσο, το ερώτημα, έτσι όπως το έθεσε ο κύριος Μέντες, είναι το εξής. Διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση για ορισμένα είδη σκαφών, ατομικά σκάφη, ότι αν δηλαδή τα αγοράσει κάποιος αλλού σε τρίτες χώρες, μετά όταν τα χρησιμοποιεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμορφούνται βεβαίως με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτή είναι μία από τις βασικότερες διευκρινήσεις ε, που μας ζητήθηκε να κάνουμε όταν συζητούσαμε ε, το νομοθετικό αυτό κείμενο. Τώρα, ως προς το θέμα του θορύβου, των επιπέδων θορύβου, είναι περίπλοκο το ζήτημα αυτό. Δεν είπαμε ότι δεν είναι εφικτό από τεχνική σκοπιά να μετρηθεί ο θόρυβο, βεβαίω και είναι εφικτό. Είπαμε ότι η αντίληψη περί θορύβου είναι δύσκολο να μετρηθεί είναι διαφορετικό ζήτημα πόσο είναι ο θόρυβος και πώς τον αντιλαμβάνεται το κοινό και μάλιστα ο καθένας από τους διαφορετικούς ανθρώπους που μπορεί να είναι παρόντες. Δεν έχουμε αναλογικό αντίκτυπο με την εισαγωγή των μέτρων μείωσης θορύβου επιβάλλοντας περαιτέρω μείωση ε, επιπέδων θορύβου που ε, ε, εκπέμπουν οι κινητήρες αυτοί. Δηλαδή, Σκοπός μας είναι να σημειωθεί πρόοδος και για να σημειωθεί πρόοδος πρέπει να ανασχεδιαστεί, να αναμορφωθεί ο κανόνας, κάτι το οποίο συνεπάγεται υψηλότατο κόστος όχι μόνο για τη βιομηχανία αλλά και για τους καταναλωτές οι οποίοι επιθυμούν να αγοράσουν κάποιο σκάφος. Οφείλουμε επιπροσθέτως να λάβουμε υπόψη το, το εξής γεγονός Ο θόρυβος έτσι όπως γίνεται αντιληπτός δεν σχετίζεται μόνο με τον κινητήρα αυτών καθ' αυτόν, αλλά εξαρτάται και, με άλλε, και από άλλες συνθήκες. Η συγκέντρωση των σκαφών, η ταχύτητα, ο καιρός. Όλοι αυτοί είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην, ε, ε, στον θόρυβο και στο, πόνο, στο πώς αυτός γίνεται αντιληπτός. Και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι διαστάσεις του ζητήματος ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να πετύχουμε ε, απτή πρόοδο. Εξού και το άρθρο 5 της ε, νομοθετικής αυτής πρότασης το οποίο άρθρο 5 δίνει τη δυνατότητα στο κράτος μέλος όπου δει όταν υπάρχει πρόβλημα φθορύβου δηλαδή, δίνεται το λόγο κρατός μέλος να υιοθετήσει μέτρα για να βρει μια ρεαλιστική ε, λύση στο πρόβλημα αυτό. Αυτά είχα να πω μέχρι αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί με τους, συνεργασία με τους ε, κατασκευαστές καφών. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα, η πρότασή σας προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να θεσπίσουν διαφορετικές εθνικές απαιτήσεις, αν θέλετε και η Επιτροπή Μεταφορών σίγουρα ενδιαφέρεται για τα θέματα αυτά ε, όπου η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να επιβάλλει ε, όρια εκπομπή θορύβων. Ενίοτε μπορεί να αξιοποιηθεί και η λύση των ε, ηλεκτρικών σκαφών όταν η εν λόγω περιοχή είναι πάρα πολύ ήσυχη και η χρήση είναι, γης είναι αμυγός αναψυχής. Εν πάση περιπτώσει, ως προς το χρονοδιάγραμμα. Θέλω να είμαστε ευέλικτοι αναλόγως με τα ευρήματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Είχα σκοπό να είχαμε ένα προσχέδιο έκθεσης ε, για τις 7 Φεβρουαρίου, μεταφρασμένο βεβαίως, το οποίο θα μας επιτρέψει να τα συζητήσουμε στα τέλη Φεβρουαρίου, 28 και 29. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 15 Μαρτίου, τις οποίες θα εξετάσουμε και θα ψηφίσουμε μετά το Πάσχα. Καλώ τους αρμόδιους συναδέλφους από τις αντίστοιχες επιτροπές που είναι αρμόδιες για τις γνωμοδοτήσεις να μας πούν αν μπορούν αυτό το χρονοδιάγραμμα να το δεχθούν και οι εν λόγω επιτροπές. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, θα μπορούσε ενδεχομένω να το ψηφίσει ε, το κείμενο αυτό στις 25 Απριλίου, εμείς στις 8 Μαΐου για να εγκριθεί από την Ολομέλεια του Ιουνίου. Αυτό το χρονοδιάγραμμα λοιπόν είναι ενδεικτικό αλλά να το συμφωνήσουμε με τους κοιόδης εισηγητές, λαμβάνοντας υπόψη ε, και την πολύ μεγάλη περίοδο που έχει περάσει κατά την προετοιμασία αυτού του και να καθυστερήσουμε ένα μήνα ή δύο μήνες δεν είναι τόσο φοβερό αφού έχουμε περάσει τόσο πολύ ε, μεγάλο χρόνο με, πάνω σε αυτό το κείμενο. Ενδεχομένως ε, μία δημόσια διαβούλευση ίσως δεν ήταν τόσο χρήσιμη. Μας ενδιαφέρει η άποψη των τελικών χρηστών αλλά και των ε, κατασκευαστών. Βεβαίως οφείλουμε να ακούσουμε και τους εκπροσώπους της ε, τοπικής αυτοδιοίκησης. Βεβαίως, ε, ε, αν υπάρχουν αρμόδια από τη Φιλανδία που θέλουν να κάνουν παρουσιάσεις, είναι ευπρόσδεκτοι για τις υδάτινες οδούς. Προχωρούμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση της κυρίας Μπάστος, την οποία καλωσορίζω. Πρόκειται για τη δική μας απάντηση στην στο έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο φυλάδιο που έχει κυκλοφορήσει για τους βασικούς 20 μίζωνες λόγους ανησυχίας των Ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων όσον αφορά στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Να, αγοράς. Να σας θυμίσω ότι εμείς το ζητήσαμε αυτό και όταν ε, δημοσιεύθηκε ε, αυτό το κείμενο, ε, ε, καλούμαστε πλέον να απαντήσουμε σε αυτό και να αντιδράσουμε. Και θα πρέπει και οι άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν από αυτού. Έχουμε καλέσει λοιπόν εκπροσώπους. Θα ακούσουμε την κυρία Μπάστος και θα συζητήσουμε μαζί της ε, την πρόοδο της έκθεσης αυτής. οι εισηγητές είναι παρόντες. Κύριος Ρέπο, ο κύριος Ροσφό δεν είναι εδώ. Η κυρία Ρούλε ε, θα απαντήσει εξ ονόματος των Πρασίνων, η κυρία Μακλάρκιν και ο κύριος Ντεγιόγκ. Κυρία Μπάστος, παρακαλώ. Ε, καλό θα ήταν να πάρετε εσείς πρώτη το λόγο για να μας ενημερώσετε για τις τελευταίες εξελίξεις. Και η κυρία Βερχόφεν είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν επικεφαλής της ειδική ομάδας για την ενιαία αγορά και το Solvent. Θα δώσω και σε εσά το λόγο για το, να μας πείτε τι στοιχεία έχετε λάβει μετά από αυτή τη δημοσίευση. Να ξεκινήσει όμως πρώτα η κυρία Μπάστος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου για να ε, κάνω την παρουσίασή μου. Θα προσπαθήσω όμως να είμαι σύντομη και περιεκτική. ως προς τους 20 μίζωνες λόγους ανησυχίας ε, Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων ε, όσον αφορά στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η έκθεση αυτή είναι ζωτικής σημασίας, πόσο μάλλον εάν αναλογιστούμε ε, τους καιρούς που διανύουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε μπροστά μας μια οικονομική, κοινωνική και χρηματοπιστωτική κρίση για πρώτη φορά στην ιστορία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ε, παρουσιάζονται κίνδυνοι ε, διάλυσης αυτού του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, κατάρρευσής του και γι' αυτό οφείλουμε να ανταποκριθούμε οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας όλες αυτές τις ανησυχίες που υπάρχουν για την ενία αγορά. Χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό εγχείρημα, χρειαζόμαστε ε, την ανοικοδόμηση της Ευρώπης η οποία θα δημιουργήσει νέες ελπίδες για τους πολίτες. Είναι αδύρυτη ανάγκη ο Ευρωπαίος πολίτης να, να τεθεί στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και βεβαίως σε αυτό το πλαίσιο συντάσσεται αυτή η έκθεση με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εντοπίζοντας τους 20 βασικούς λόγους, τα 20 βασικά προβλήματα από πλευράς Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων ως προς τη λειτουργία της ενέας αγοράς. Οι πολίτες ταξιδεύουν, οι πολίτες ε, κάνουν... Ε, μεταβαίνουν από τη μία χώρα στην άλλη για να εργαστούν, για να ζήσουν Επιχειρήσεις επίσης θέλουν και να εγκατασταθούν και εγκαθίστανται αλλού στην Ευρώπη. Είναι ένα πρόβλημα δηλαδή που έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητα. Τίθενται λοιπόν διάφορα ζητήματα εκεί. Υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας, θέματα κατοικίας, άδεια παραμονής. Ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες που εγκαθίσταται σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, αναγνώριση των προσόντων τους, μη διάκριση ε, ως προς τις ευκαιρίες απασχόλησης, ε, πρόβλημα καταχώρησης των πινακίδων των οχημάτων, ε, πρόβλημα αναγνώρισης διπλωμάτων και πτυχίων. Θα μπορούσα να επεκταθώ ιδιαιτέρως σε κάθε έναν από αυτούς τους 20 μείζονες λόγους. Θέλω όμως να είμαι σύντομη και περιεκτική. Η έκθεση αυτή προσφέρει μια συνολική θεώρηση των εμποδίων στα οποία προσκρούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Η έκθεση κάνει μια ανάλυση βάσει των στοιχείων που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε το δίκτυο Solvit, έχουμε το Enterprise Europe Network, τις ενώσεις καταναλωτών, τα σημεία επαφής για να μην μακρηγορήσω. Έχουμε βασίσει την έρευνά μας σε πολλές και διαφορετικές πηγές. Επομένως, τρία είναι τα βασικά κενά που πλήττουν την ενιαία αγορά και που σχετίζονται με την πληροφόρηση. Διαπιστώνουμε καταρχάς κενό πληροφόρησης, πολύ μεγάλο. Πολύ συχνά οι πολίτες είτε δεν γνωρίζουν είτε δεν κατανοούν πλήρως τα δικαιώματά τους, δεν γνωρίζουν πού μπορούν να βρουν τις πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν. Δεύτερο κενό που έχουμε διαπιστώσει είναι το κενό εφαρμογής ε, θέση σε ισχύ του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πάρα πολλούς τομείς υπάρχει χάσμα μεταξύ νομικού πλαισίου που έχει τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τρόπου εφαρμογής της νομοθεσίας στην πράξη. Άλλωστε, ε, δημιουργείται, έχει δημιουργηθεί ένα νομοθετικό κενό κάτι το οποίο δείχνει ότι το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών και επιχειρήσεων. Πολύ συχνά όλα αυτά σχετίζονται με το γεγονός ότι κατά την άποψη του πολίτη η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να γνωρίζει και να ρυθμίζει συγκεκριμένους τομείς ενώ αρμοδιότητα έχει το κράτος μέλος ή αντίστροφα. Έχουμε τις τρεις ελευθερίες, ε, το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης, πράγματα δηλαδή που πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα, δεδομένης μάλιστα και της ε, περίοδου ε, την οποία διανύουμε αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό μας οικοδόμημα. Είναι ένα τεράστιο κεκτημένο του ευρωπαϊκού γίγνεσθε και θα πρέπει να υλοποιείται και να εφαρμόζεται κάθε μέρα στην πράξη. Και ο Επίτροπος Μπαχνιέ άλλωστε, ο οποίος είναι ο αρμόδιος Επίτροπος, το έχει τονίσει επανειλημμένος. Είναι δική μας ύψιστη υποχρέωση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ανταποκριθούμε και να προσφέρουμε λύσεις σε αυτά τα 20 προβλήματα τα οποία είναι τα 20 πρώτα στον πολύ μακροσκελή κατάλογο προβλημάτων. Καλό είναι ότι έχουμε ήδη υιοθετήσει μια κάποια προσέγγιση και ήδη υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δύναται να ανταποκριθεί τροποντινά. Λοιπόν, πολύ συχνά τα κράτη-μέλη μας δεν εφαρμόζουν με επιμέλεια το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Στην ενσωμάτωση των οδηγιών και λοιπόν διατάξεων χάνονται κάποιες λέξεις στην πορεία. Δεν τηρούνται με αυστηρότητα όλες αυτές οι προθεσμίες που πρέπει για να διευκολυνθεί η ζωή των φοιτητών, των πολιτών, των ταξιδιωτών, των εργαζομένων. Για να διευκολυνθεί επίσης η λειτουργία των επιχειρήσεων σε αυτό τον ευρωπαϊκό ε, κοινό χώρο που μας ανήκει. Σήμερα, σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οφείλουμε να διευκολύνουμε την την κινητικότητα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Οφείλουμε να είμαστε διατεθειμένοι να διαδραματίσουμε τον οικονομικό, κοινωνικό και εμπορικό ρόλο που μας αναλογεί ε, στην ε, ε, παγκοσμιοποιημένη οικονομία αυτή τη στιγμή. Εάν σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, θα μπορέσουμε να καταλαγιάσουμε τις καθημερινές ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών. Εάν καταφέρουμε να δώσουμε ικανοποιητικές απαντήσεις, σίγουρα θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του Ευρωπαίου πολίτη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Είναι δικό μας καθήκον η έκθεση αυτή έχει τεράστια συμβολική αξία πέραν όλων των άλλων και δίνει, προσπαθεί να δώσει μια ταχεία αποτελεσματική λύση ε, ούτως ώστε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις προκλήσεις που υψώνονται μπροστά μας. Ούτως ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Πιστεύω ακραδάντως ότι είναι μια έκθεση πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ σημαντική. Ε, χαιρετίζω τους σκιώδεις εισηγητές, εκφράζω την ελπίδα μου για μια αγαστή συνεργασία μεταξύ μας και ελπίζω και οι οκτώ επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες θα συμμετάσχουν στην ε, ε, κατάρτιση της τελικής έκθεσης να συμβάλλουν Επιτροπή Πολιτισμού, Οικονομίας, Απασχόλησης, Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Νοεμικών Θεμάτων, ε, Μεταφορών μεταξύ άλλων. πολλές και διαφορετικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ε, κληθούν να συμμετάσχουν. Είναι ένα πολύ κοπιώδες έργο αυτό. Ωστόσο, θα αποφέρει καρπούς και έτσι θα εκπέμψουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς τον Ευρωπαίο πολίτη. Θα ήθελα να ολοκληρώσω κάπου εδώ την παρέμβασή μου για να υπάρξει χρόνος και για συζήτηση. Ε, περιμένω, ε, με αδειμονώ να ακούσω τις απόψεις των σκιωδών εισηγητών και θα ήθελα να πω ότι θα προχωρήσουμε από τις 19 μέχρι 21 Μαρτίου, μετά τροπολογίες μέχρι τις 12 Απριλίου, αξιολόγηση τροπολογιών στις 8 Μαΐου και ε, ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή 19 Ιουνίου και έγκριση στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Αυτά ως προς το χρονοδιάγραμμα. Βεβαίως έχουμε μία συμφωνία για τα σημεία 7 και 12 τα οποία έχουν να κάνουν με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, το 7 μεν και το 12 για την πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από πλευράς πολιτών και θα πρέπει να οριστεί ξεκάθαρα η αρμοδιότητα και ποια θα είναι η ιεράρχηση ε, μεταξύ των διαφόρων επιτροπών. Αυτά προς το παρόν ε, παραμένω στη διάθεσή σας, δεν θα πω τίποτα άλλο ε, αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Μπάστος, λέει ο Πρόεδρος. Χαίρομαι διότι συνεργάζεστε με τις άλλες επιτροπές και περιμένουμε να δούμε τη δική τους πρόοδο. Λοιπόν, βλέπω ότι ο κύριος Ρέπο είναι ο κύριος ε, Σκιώδης που είναι παρόν. Ο κύριος Μάντερς θα ε, μιλήσει εξ ονόματος του κύριου Ροσφουκό που είναι απόν. Καλωσορίζω ε, τον κύριο Ντεγιόν, την κυρία ε, Εσείς είστε σκιώδης εισηγητής ή εισηγητής για μια άλλη επιτροπή. Ναι, η απάντηση εκτός μικροφώνου δυστυχώς. Πολύ καλά λέει ο πρόεδρος και η κυρία Γκέπχαρτ. Επομένως, αυτός είναι ο κατάλογος ομιλητών. Να ξεκινήσω με τον κύριο Ρέπο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ εύκολο να εκφράσω την πλήρη μου συμφωνία με τις απόψεις που εξέφρασε η κυρία Μπάστος. Έχει φανεί ξεκάθαρα ότι η εσωτερική αγορά έχει ευεργετική επίδραση και στους Ευρωπαίους πολίτες και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Και αυτό το διαπιστώνουμε τα τελευταία 20 χρόνια. Ωστόσο, για πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαντάζουν ε, ξένα προς αυτόν. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να πείσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τα ωφέλη της εσωτερικής αγοράς. Προσωπικός. Ε, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το ζήτημα της κοινοτικότητας των εργαζομένων και των επαγγελματικών προσόντων και της αναγνώρισης αυτών. Θα πρέπει να αρθούν όλα τα εμπόδια που έχουν να κάνουν με το ηλεκτρονικό εμπόριο επίσης. Οφείλουμε να αναζητήσουμε μέσα που θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια. Επίσης, η αρχή της ε, εθελούσιας βάσης της εθελοντικής συμμετοχής στην επίλυση των διαφορών. Όλα αυτά είναι πρακτικές ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα πρέπει να τις εξελίξουμε έτσι περαιτέρω. Είναι όλα αυτά πολύ σημαντικά για τους οικονομικούς φορείς, ούτως ώστε να αποφευχθούν ε, να, τα δικαστήρια και να υπάρχει εξοδικαστική επίλυση των διαφορών. Από εκεί και πέρα έχουμε και το πρόβλημα της δραστηριότητας ή της απραξίας των εθνικών αρχών. Πάρα πολύ συχνά η υλοποίηση, η εφαρμογή μιας οδηγίας ή ενός νομοθετικού κειμένου εν γέννη ε, ήταν αρκετά προβληματική και πολύ συχνά υπέστησαν αδικίες οι Ευρωπαίοι πολίτες κατά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κάτι το οποίο δείχνει ότι δεν έχουν πάντοτε οι Ευρωπαίοι πολίτες όλες τις ευκαιρίες που θα έπρεπε και δεν επιδεικνύουν πάντοτε τα κράτη-μέλη τη βούληση να συμμορφωθούν ε, με τα συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν έχει κανένα νόημα ότι έχει συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο εάν δεν εφαρμόζεται στην πράξη καθημερινά σε εθνικό επίπεδο. Και αυτές είναι οι βασικές σκέψεις που θα ήθελα να εκφράσω. Οφείλουμε λοιπόν να στηρίξουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, να διευρύνουμε τις δυνατότητές τους και να στηρίξουμε και τις εθνικές αρχές για να γνωρίσουν καλύτερα ε, τους διάφορους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Σε βάθος, χρόνο, σε βάθος χρόνου αυτό θα ωφελήσει εξαιρετικά την ενιαία εσωτερική αγορά. Υπό την διεύθυνση της κυρίας Μπάστος θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή έκθεση για να προωθήσουμε την εσωτερική αγορά και να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μάντερς. Α, ωραία. Κυρία Ρούλα. Ο κύριος Ντιγιόγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να παρατηρήσω ότι κατά την άποψή μου υπάρχουν τρεις κατηγορίες προβλημάτων. Υπάρχουν βασικά προβλήματα πρώτα-πρώτα. Άμα ε, κάνω μια κουβέντα για την εσωτερική αγορά στην πατρίδα μου, στο σπίτι μου ε, αναγκάζομαι να μιλώ πάρα πολλές ώρες για να εξηγήσω τι είναι η εσωτερική αγορά δεν έχω πρόβλημα αλλά αυτό ε, δείχνει το πώς κατανοεί ο Ευρωπαίος πολίτης στην ευρωπαϊκή αγορά. Μιλώ για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, για τα εργασιακά προβλήματα και, και τα λοιπά και τα Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στην Πορτογαλία και στην... από την Πορτογαλία και την Ελλάδα να μετακομίζουν πολλές επιχειρήσεις στην Ολλανδία όχι γιατί αισθάνονται πιο καλά ή έχει καλύτερο καιρό προφανώς αλλά γιατί είναι το φορολογικό ε, καθεστώς πιο ευνοϊκό για αυτούς. Είναι ε, ε, σκανδαλώδες αυτό και ο κύριος Μόντι αναφέρθηκε σε αυτό αν δεν κάνω λάθος λοιπόν θα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε κάτι τέτοια πράγματα. Η επαφή με, το κοινό, με τους πολίτες μας, με την κοινή γνώμη είναι πολύ σημαντική και στις επαφές που έχουμε θα πρέπει όχι να ασχολούμεθα με τεχνικά θέματα που ενδεχομένως δεν ενδιαφέρουν και πάρα πολλούς αλλά να ε, μιλούμε για γενικότερα θέματα σαν και αυτό που σας είπα μόλις πριν από λίγο. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν ε, και άλλα ζητήματα το roaming ας πούμε είναι κάτι που άγγιξε τους πολίτες και το θέμα της ενέργειας προσφορές στην αγορά ενέργειας που είναι πολύ περίπλοκο θέμα και οι καταναλωτές παραπονιούνται γι' αυτό θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό στην Επιτροπή αυτή. Στη δεκαετία του 90 θυμάμαι ότι προσπάθησα να χρησιμοποιήσω μια πιστοτική κάρτα στη, ε, στο Βέλγιο, η οποία πρέπει να πληρωθεί στην Ολλανδία. Δεν είχε καθόλου τίποτα να κάνει με την νέα και εύρυθμα λειτουργούσα ε, ευρωπαϊκή αγορά. Κάθε άλλο. Δεν σα περιγράφω τα προβλήματα που έχω και τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν. διαφορετικό ΦΠΑ είναι δύσκολο και για του επιχειρηματίε αλλά και για του κοινού θνητή να αντιμετωπίσουν το θέμα. Είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και βέβαια, βέβαια είναι και διάτριτο και ε, ευάλωτο σε οποιαδήποτε απάτη. Τι άλλο, οι πωλήσει μέσω μέσω ίντερνετ. Πολύ σωστά αναφέρθηκε. Αυτό είναι όντω αυτή η διεύθυνση και η πορεία θα κάνουμε στο μέλλον. Θα πρέπει να είναι πραγματικά υποχρεωτικό να δημιουργηθεί κάποιο πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα και ότι οι πωλήσει μέσω ε, διαδικτύου θα είναι πραγματικά ασφαλεί και θα προστατεύεται το τοπίο αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να καλυφθούν εδώ και δίνω όλε τι καλύτερε ευχέ μου στην ε, εισηγήτρια για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να πραγματευτεί όλα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα μαζί σας με την ανάγκη να αντιμετωπιστούν κάποια από τα δύσκολα αυτά θέματα που κάνουν δύσκολη τη ζωή των πολιτών. Γιατί αυτό το θέμα της ενιαίας αγοράς μπορεί ζητείται εδώ και χρόνια και ποτέ θα το έχουμε πετύχει εδώ και χρόνια, αλλά εν τούτης ακόμα τίποτα δεν έχει γίνει. Κύριε Κιούι καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έγγραφο εργασίας, το οποίο είναι πάρα πολύ καλά δομημένο και προσωπεύει μια νέα προσέγγιση, η οποία θέτει τις σωστές διευθύνσεις για την μελλοντική εργασία μας. Ε, ασπάζομαι πλήρως και συμφωνώ με την πρώτη ιδέα που αναφέρεται στο έγγραφο αυτό, ότι δηλαδή η εσωτερική αγορά είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτεύξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά οι προσδοκίες εκ μέρους των πολιτών είναι επίσης πάρα πολύ ψηλές και πρέπει να μπορέσουμε να αποκριθούμε με σαφήνεια και χωρίς καμία αμφισημία απέναντι στους πολίτες σε σχέση με τα ερωτήματα και τις καταγγελίες τους. Και αυτό ιδιαίτερα μετά την χρηματοπιστωτική κρίση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να θεωρήσουμε και να ξαναδούμε το θέμα των ε, εσωτερικού μηχανισμού της αγοράς. Ελπίζει σημαντικό και ευπρόσδεκτο στο έγγραφο εργασίας και στην έκθεση είναι ότι παίρνουμε κάποια απόσταση και κοιτούμε την λειτουργία του συνόλου της εταιρική αγοράς. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο. Αυτού θα ήθελα ιδιαίτερα να εστιάσω σε δύο θέματα, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται στο συνολικό έγγραφο, αν και εκτιμώ ιδιαίτερα την ευκαιρία που έχω λειτουργώντας ε, ως ε, αναπληρωτής ε, στην Επιτροπή αυτή. Εκπροσωπώ επίσης την κύρια Επιτροπή στην οποία εργάζομαι και ως εκ τούτου θα ήθελα καταρχάς να επικεντρωθώ στα θέματα ενέργειας και μεταφορών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής, στην οποία είμαι πλήρε μέλλον. Σε σχέση τώρα με την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες, ευχαριστώ την προσοχή σας στις ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε τους δύο τομείς. Σε ό,τι, τομείς. Σε ό,τι αφορά τις ε, ομοιότητες, δυστυχώς αναδύεται το ερώτημα της έλλειψης εφαρμογής του υφιστάμενου νομικού πλαισίου στα εθνικά δίκαια. Και αυτό ισχύει για μια σειρά κρατών μελών. Στο πεδίο της ενέργειας, 18 κράτη-μέλη υπόκεινται και έχουν παραπεμφθεί λόγω της μη εφαρμογής. Ο ακριβής αριθμός είναι 16 στο πεδίο το αντίστοιχο αριθμό είναι 16 κράτη-μέλη στο πεδίο τηλεπικοινωνιών. Και αυτό μα εμποδίζει βέβαια να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο τη σχετική κοινοτική νομοθεσία στο θέμα αυτό, γιατί δεν έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή και δεν έχει μεταφερθεί στα εθνικά δίκαια όλων των κρατών μελών. Και σε ό,τι αφορά τι διαφορέ των δύο αυτών πεδίων από τη σκοπιά του καταναλωτή, Το σημαντικό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές στον τομέα ενέργειας, ενώ τα αντίτυπα και οι τιμές στις τηλεπικοινωνίες μπορεί να μην έχουν πέσει δραματικά, αλλά πάντως έχουν μειωθεί. Πιστεύω ότι σε σχέση με τον τομέα ενέργειας, η αύξηση των τιμών οφείλεται καταρχάς στις αυξήσεις των πρώτων υλών. Και αυτό το οποίο δεν μπορέσαμε να επιτύχουμε σε ό,τι στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας είναι ότι δεν καταφέραμε να, με την ομοθεσία μας να προστατεύσουμε πραγματικά τους καταναλωτές. Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα στο τομέα της ενέργειας γιατί η, η, η διάρθρωση των τιμολογίων κατά βάση διευθετείται ή είναι ακόμα κεντρικά κατευθυνόμενη και δεν υπάρχει σχετική διαφάνεια. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να ερμηνεύσουμε, ο καθημερινός καταναλωτής να ερμηνεύσει ακριβώς τη τιμολογία. Βρίσκουν όλοι τους ε, λογαριασμούς ε, του ηλεκτρικού εξαιρετικά πολύπλοκους και πάρα πολλά πρέπει να γίνει στο πεδίο αυτό, αν και τα περισσότερα προβλήματα συνδέονται με θέματα υποδομής. Ε, επιτρέψτε να αναφέρω σχετικά τα εφή δίκτυα ή την εισαγωγή των εφιών μετρητών. Ερχόμενοι τώρα στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών, οι τιμές μειώνονται σταθερά, αν και θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο και λανθασμένο να καταλήξουμε σε τελικά αποτελέσματα σχετικά. Παρά την πτώση των τιμών, οι μηχανισμοί της αγοράς δεν λειτουργούν σωστά. Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι χειριστές δεν δίνουν σαφείς προφορίες σχετικά με τα προϊόντα τους, τις υπηρεσίες τους και τα πακέτα τα οποία παρέχουν. Και τα περισσότερες από τις καταγγελίες των καταναλωτών ακριβώς αναφέρουν το πρόβλημα αυτό. Είμαι πεπισμένος ότι η εμπειρία την οποία έχουμε και την οποία θα κερδίσουμε στο πεδίο της περιαγωγής, του roaming, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε, και σε ευρύτερο πεδίο. Δεν θέλω να προικάσω και να προδικάσω αποτελέσματα, γιατί θα έχουμε αρκετό χρόνο να εργαστούμε συλλογικά. Αλλά κάποια πρώτα συμπεράσματα στα παιδιά αυτά και σε άλλους τομείς που καλύπτονται από τα 20 ερωτήματα, νομίζω ότι τελικά η έκθεσή μας δεν θα είναι ισμάτη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε και μιλήσατε για τα κρίσιμα αυτά ζητήματα. Συμφωνώ μαζί σας ότι ακριβώς ε, οι εθνικοί πάροχοι, ιδιαίτερα στη ενέργεια, θα πρέπει να συντονιστούν καλύτερα για να αντιμετωπίσουν αυτά τα πολύπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές σε μια απελευθερωμένη αγορά. Και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε σχετικές ιδέες για μια χάρτα των καταναλωτών. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία για την Επιτροπή μας, κατά προστασία του καταναλωτή, να παρουσιάσει και να κάνει την συνεισφορά της. Ευχαριστούμε και τις δικές σας προτάσεις. Κυρία Κέπα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπάστος για την παρουσίασή της και για την... Ε, τις εξηγήσεις που έδωσε. Αλλά όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι και εγώ έχω ε, πρόβλημα στην πατρίδα μου να εξηγήσω στους ε, συμπολίτε μου ότι η εσωτερική αγορά είναι καλό πράγμα. Οι, οι πολίτες ε, συνεχώς μιλάνε για τις Βρυξέλλες κοίτα τι κάνανε οι Βρυξέλλες όλα τα αποφασίζουν οι Βρυξέλλες δεν είναι έτσι η, αυτό νομίζω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι δεν παρουσιάζουμε αρκετά ε, έντονα τα θετικά πράγματα που κάναμε για τους πολίτες. Άρα αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει από όλους μας και με μεγαλύτερη ένταση. Βεβαίως ξεκινήσαμε ε, για τα θέματα της εσωτερικής αγοράς και της προστασία του καταναλωτή από τα 20 παλιά αιτήματα αν θέλετε που υποτίθεται ότι είχαν οι Ευρωπαίοι πολίτες κτλ. Και, ε, και πού φτάσαμε. Κοιτάξτε, όταν ακούμε νεαρούς που λένε ότι ήθελα να ανοίξω λογαριασμό στην τράπεζα και δεν μπορούσα να ανοίξω λογαριασμό γιατί δεν είχα μια διεύθυνση στην οποία διαμένω μονίμως και βεβαίως δεν μπορούσα να πιάσω σπίτι γιατί δεν είχα λογαριασμό στην τράπεζα αυτή είναι η Ευρώπη που προσφέρουμε στους νέους δεν είναι η καλύτερη εμπειρία αυτή για ένα νέο όταν μου πει ένας α, ένα άτομο με αναπηρία ξέρεις πήγα στη Φραγκφούρτη και το λέω γιατί είναι ο τόπος μου Φραγκφούρτη και παρόλο που ήμουνα στη, σε θέση αναπήρων την οποία δικαιούμαι να πάω βάσει του δικού μου, βάσει του ενός χαρτιού που έχω, ε, πήρα κλίση διότι δεν αναγνωρίστηκε το πιστοποιητικό που έχω, γιατί δεν προέρχεται από το Δήμο Φραγκφούρτης. Λοιπόν, δεν είναι δυνατό να τα δεχόμαστε αυτά. Επίσης, στο εξωτερικό, πάμε στο εξωτερικό, τηλεφωνούμε και παρά τις προσπάθειες που έγιναν στο roaming, ε, ε, πληρώνουμε πάρα πολλά δεν επιτυχάνει το roaming, δεν γίνεται το roaming θέλουμε να κάνουμε και και και χίλια δυο καθημερινά παραδείγματα θα μπορούσα να σας αναφέρω αυτή λοιπόν είναι η ανησυχία που έχουμε οι ανησυχίε που είχαν ανέκαθεν οι Ευρωπαίοι πολίτες υπάρχουν προβλήματα δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ότι είναι εύκολο να λυθούν αλλά θα πρέπει να αγωνιστούμε για να βρούμε τις λύσεις με αυτή την έκθεση της κυρία βάστως είναι πάρα πολύ σημαντική και πολύ σημαντική και από πολιτική άποψη διότι απευθύνεται ασχολείται με την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και βεβαίως ε, αυτό πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα να διευκολύνουμε την καθημερινή ζωή του πολίτη να επέμβουμε εκεί. Γι' αυτό ευχαριστώ την κυρία Μπάστος για την έκθεσή της, τη συγχαίρω για το πώς παρουσιάζει τα πράγματα και ελπίζω να καταλήξουμε, είμαι σίγουρη μάλλον θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή γνωμοδότηση την οποία θα καταλάβουν και θα αναγνωρίσουν. Είμαι σίγουρη και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Πολύ για τα σχόλια αυτά. Ίσως κάποια καταληκτήρια σχόλια και να προσκαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, κάνει, να δώσει τα αντίστοιχα καταληκτήρια συμπεράσματα και κάποιες ιδέες. Ίσως την απάντηση της κυρίας Φόβενον από τη διάφορα σχόλια των μελών της Επιτροπής. Απλώς επιτρέψτε μου να πω ότι αξίζει να, να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η δημοσίευση της έκθεσης και τα ευρήματά της δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο φόρουμ της ενιαίας αγοράς, το οποίο παρακολουθήσαμε πολύ εξημών στην Κρακοβία και υπήρχαν κάπου 5.000 άτομα από όλη την Ευρώπη που παρακολούθησαν το φόρουμ αυτό και από πολλούς διαφορετικούς τομείς της ε, οικονομίας και ήταν φοιτητέ, νεαροί, ε, ε, άνθρωποι, επαγγελματίες, ακόμα και σταξιούχοι. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση αυτή και είχαμε πάρα πολύ feedback από το φόρουμ αυτό και κάποιες από τις ανησυχίες των καταναλωτών. Ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι ότι οι λύσεις σε πολλά από τα ζητήματα τα οποία ε, εγείρουν οι, οι, οι πολίτες πρέπει να αντιμετωπιστούν σε σχέση με τις εθνικές αρχές. Όπως για παράδειγμα η, η οι πινακίδες κυκλοφορίας η πρώτη, για πρώτη φορά ένταξη αυτοκινήτων ή και θέματα οικογενειών, όταν έχουμε μάλιστα μικτούς γάμους. Κάποια θέματα τα οποία εθίγησαν στην έκθεση του κυρίου Λαμασούχ που υπέβαλε στον κύριο Σαρκοζή πριν από τέσσερα χρόνια, καθόλου δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Ελπίζω ότι με την έκθεση αυτή και συνεισφέροντας και από άλλες επιτροπές μπορεί ίσως να ανεβάσουμε το πολιτικό προφίλ, του θέματος και να αναλυφθεί κάποια δράση. Γιατί είναι σαφές ε, ότι η λαϊκή συμμετοχή για την ε, ενιαία αγορά δεν είναι τόσο ισχυρή όσο ήταν, γιατί πλέον στις περιλές περιπτώσεις το βλέπουμε περισσότερο σαν απειλή παρά σαν ευκαιρία. Γιατί έχουν δημιουργηθεί σχετικές αρνητικές ε, εντυπώσεις για τις, λόγω της πολύ μεγάλων ασυνεπιών της ενιαίας αυτής αγοράς. Και ιδιαίτερα η αγορά online αγορών που εθίγει, όπου πολίτες οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν online και είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση και αγοράση υπηρεσιών ή, υπηρεσιών ή προϊόντων που θεωρούν ότι δικαιούνται και έχουν το, δικαιούνται να έχουν, δεν μπορούν να το κάνουν. Ήταν απόλυτα σωστό να προσκαλέσουμε τους συναδέλφους στο Κοινοβούλιο και να κάνουμε εμείς οι ίδιοι την άσκηση αυτή. Γιατί δεν έχει νόημα να πιέζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τη δουλειά αυτή. Γιατί αν μένει αυτή η εργασία και αυτή η έκθεση στο ράφι και κανείς δεν παρακολουθεί τα επιγενόμενα, δεν έχει κανένα νόημα. Γι' αυτό ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πιο δομημένη και ε, πιο επιμελή παρακολούθηση της έκθεσης που έχει συντάξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δική μου, αν θέλετε, αντίδραση εν μέρη απηχεί και την άλλη Επιτροπή της οποίας ε, υφίσταμε. Κύριε Χαβελχόβεν, έχετε κάτι να πείτε. Ένα σύντομο σχόλιο. Καταρχάς, ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί με δική σα πρωτοβουλία απολαύσαμε ιδιαίτερα την εκπόνηση εργασία αυτής. Και επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοούμε τη σημασία της εργασίας αυτής. Σε ό,τι αφορά την απόκριση μέχρι στιγμή από πρακτική σκοπιά, πρέπει να πω ότι κατά κάποιο τρόπο έχει γίνει ένα best seller. Μα ζητείτε συνέχεια να κάνουμε αντίγραφα τη έκθεση αυτή και να το στέλνουμε σε όλε τι γωνιές τη Ευρώπη. Επομένω, συζητείται η έκθεση αυτή όχι μόνο σε ευρωπαϊκά φόρα, αλλά και εθνικά φόρα, όπου εκεί πρέπει να γίνεται ακριβώ η συζήτηση. Άρα ήδη εκπληρεί του σκοπού τη η, έκθεση, η μελέτη αυτή. Εξάλλου, σε ό,τι αφορά τον απόκριση στο δικό μου επίπεδο, μπορώ να πω ότι αν μη τι άλλο υπάρχει όλο και μεγαλύτερη προσοχή ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν τα χάσματα αυτά και τα τρία ταυτόχρονα. Όχι μόνο περισσότερη νομοθεσία, αλλά ταυτόχρονα πληροφόρηση και επίσης σωστή εφαρμογή όλων των θεσπιζόμενων κανόνων. Αυτό είναι κάτι που επίσης έχει βοηθήσει η έκθεση αυτή να δημιουργήσει ε, όλο και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση και βλέπουμε ότι στην Επιτροπή και πάρα πολλοί έχουν πάρει σοβαρά το θέμα αυτό. Αυτό επηρεάζει λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται και εκπονούν λύσεις. Αλλά όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, πρέπει να το κάνουμε μαζί με τους ε, βασικούς παίκτες αγοράς. Αυτό ήθελα να πω σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ. Και προσβλέπουμε στην περαιτέρω συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να σας ζητήσω ο σχεδιασμός σας από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει κάποια σύνοψη, αν θέλετε, των σχετικών αποκρίσεων, κάποιο σχετικό πρόγραμμα, γιατί οι δείκτες συζητώνται παντού. Υπάρχει κάποιος μηχανισμός συλλογής των ε, απαντήσεων. Όχι, μέχρι στιγμής όχι γιατί ακριβώς δεν έχουμε λάβει και όλες τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια. Όταν στείλαμε τα φυλάδια για γεγονότα και εκδηλώσει σε εθνικό επίπεδο, δεν ξέρουμε ποιο είναι ο αντίκτυπος της όλης συζήτηση, συζήτησης σε επίπεδο κράτους μέλους. Δυστυχώ μέχρι στιγμή δεν υπάρχει σχετικό μηχανισμός που να καταγράφει τι αντιδράσει κυρία Μπέστος ίσως θα πρέπει να το εξετάσει αυτό. Θέλετε να μας πείτε πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα και οποιοδήποτε άλλο σχετικά θέματα ή σχόλια τα οποία θέλετε να κάνετε σχέση με αυτά που ακούστηκαν εδώ στην Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ όλα τα μέλη της ε, Επιτροπής που συνεισέφεραν στην όλη συζήτηση. πρέπει να γίνει η κάλυψη των τριών αυτών κενών, που δεν είναι κάτι καινούριο. Η έκθεση δημόνων το 1995 ήδη εντοπίζουν αυτά τα κένα. Χάσμα στην πληροφόρηση και μη εφαρμογή των σχετικών οδηγιών και διαπιστών και ένα νομικό κενό. Έχει γίνει λοιπόν η διάγνωση, πρέπει πλέον να δράσουμε πρέπει να αναλυφθεί δράση για να καλύψουμε αυτά τα κέννη. και αυτό πρέπει να γίνει ταυτοχρόνως. Διαφορετικά, εάν, κάνουμε, εάν παρέμβουμε μόνο στο θέμα της πληροφόρησης ή μόνο της εκπόνησης νέων οδηγιών, ή αν μείνουμε μόνο στην νομοθεσία περαιτέρω εμβάθυνση του ευρωπαϊκού έργου με καινούργια νομοθεσία χωρίς να παρακολουθούμε μια ταυτόχρονη και ολοκληρωμένη προσέγγιση και στα τρία μέτωπα, τότε οι πολίτες θα συνεχίζουν να μην καλύπτονται και να μην εισακούονται. Αυτό που ελέγχθη λοιπόν είναι πολύ σωστό, είναι πολιτικό το ζήτημα. Πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση ε, ανταπόκρισης και βελτίωσης και θα πρέπει να εμπλακούν οι εθνικές αρχές προκειμένου να καταφέρουμε να απαντήσουμε στις θεμελιώδεις αυτές ανησυχίες των πολιτών. Εάν γίνει αυτό, θα έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα στην, στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την, την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το θέμα συγκεκριμένα, το οποίο αν θέλετε άπτεται των πολύ μεγάλων ανησυχιών που εντοπίζουν επιχειρηματίες και πολίτες, αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, την ενέργεια, την εισαγωγή οχημάτων, το προβλήμα το οποίο αντιμετωπίζουν οι φοιτητέ. Και ανοίγω μικρή παρένθεση για να πω ότι ένας φοιτητή που έρχεται από ένα κράτος μέλος για να κάνει σε ανταλλαγή, στα πλαίσια ανταλλαγή φοιτητών στο πρόγραμμα Εράσμους αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα τα οποία σαφέστατα εντοπίστηκαν από τους, αυτούς που έκαναν την έρευνα φτάνουν στο κράτος μέλος πρέπει να ανοίξουν ένα λογαριασμό στην τράπεζα γιατί ο ιδιοκτήτης ε, του διαμερίσματος το οποίο θα ενοικιάσει το απαιτεί εμφανίζεται στην τράπεζα να ανοίξει το λογαριασμό φοιτητή, αλλά από πλευρά τη η τράπεζα απαιτεί να υπάρχει κάποιο έγγραφο είτε ότι έχει κάρτα παραμονή είτε μια απόδειξη εργασία. Όμω ο φοιτητή δεν έχει να εργαστεί, ούτε έχει σύμβαση εργασία, ούτε έχει και τίτλο παραμονής, γιατί δεν έχει ακόμα ενοικιαστήριο. Ιδού ένα παράδειγμα συγκεκριμένο του φαύλου κύκλου και των καθημερινών διδασκαλίων δυσκολιών που δυσκολεύουν την κινητικότητα των ε, πολιτών στον ε, κοινό μας ευρωπαϊκό χώρο. Εξάλλου, για τα υπόλοιπα σημεία, όλα τα οποία εντοπίστηκαν είναι ζωτική σημασία. Η ενέργεια, η προάσπιση των συμφερών των καταναλωτών, στην επιλογή σε επιλογή τους απέναντι στους παρόχους ενέργειας. Ιδού άλλο ένα ζήτημα το οποίο αφορά στο συντονισμό και εθνικής νομοθεσίας, όπως πολύ σωστά είπε ο Πρόεδρος, και κυρίως εξαρτάται από την βούληση, την πολιτική βούληση των κυβερνήσεων των κρατών μελών και βέβαια αυτό αφορά και στην εναρμόνιση η οποία απαιτείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδού οι ανησυχίες οι οποίες ε, έχουν καταγραφεί με σαφέστατο τρόπο, είναι πολύ καλά στοχευμένες, έχουν εκφραστεί από τους πολίτες και είναι ζητήματα τα οποία και εμείς α, εντοπίζουμε ως και θεωρούμε και χαρακτηρίζουμε πολύ μεγάλα εμπόδια για την πραγματική υλοποίηση της ενιαίας εσωτερική αγοράς. Επιπροσθέτως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν έρχονται εδώ και παραπονούνται και λένε ότι, ε, πρέπει, ότι είναι πραγματικά η ραχοκαλιά της ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης και η ατμομηχανή τη ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζουν τεράστιε όμω δυσκολίε που εμποδίζουν την επέκτασή του πέραν των εθνικών ορίων στην ενιαία εσωτερική αγορά πέρα δηλαδή από την χώρα έδρας, αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες αυτές ενώ ο καθένας γνωρίζει ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση ανεργίας και γνωρίζουμε ότι το 90% των θέσεων απασχόλησης παρέχεται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ιδού λοιπόν οι απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε και αντιμετώπιση ταυτόχρονα σε τρία αυτά πεδία που έχουν αντιμετωπιστεί και έχουν εντοπιστεί εδώ και πάνω από δεκαετία είναι θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με την ζωηρή και στεναρή εμπλοκή και των θεσμικών οργάνων και των εθνικών κρατών μελών. Το χρονοδιάγραμμα το οποίο προβλέπεται μας δίνει τον χρόνο στοχασμού και εργασίας πάνω στα θέματα αυτό, εργασίας ε, εις βάθος και με λεπτομερή τρόπο, το έλεγα προηγουμένως, έδωσα τις ημερομηνίε. Το Μάρτιο ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή, εδώ δηλαδή, τη δική Επιτροπή. Στη συνέχεια το χρονοδιάγραμμα προβλέπει κατάθεση, συγγνώμη, 2 Απριλίου ε, προθεσμία για υποβολή προτάσεων, Μάιο ε, στη, στο Κοινοβούλιο συζήτηση και τελική συζήτηση την Ολομέλεια του Σεπτέμβριο. Ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο μας δίνει το χρόνο συζήτησης να υπάρξει ε, αλληλοπαράθεση επιχειρημάτων και έχουμε επίσης τον χρόνο που μας, επιτρέπεται να έχουμε και ακροάσεις ήδη μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Επιτροπή εδώ για να ανοίξουμε το θέμα αυτό, για να δημιουργήσουμε πραγματικά ένα μέτωπο έλεγα ότι προβλέπεται την επόμενη εβδομάδα συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσουμε με πιο στοχευμένο τρόπο το ζήτημα. Έχω την πρόθεση να ξεκινήσω από τώρα να εργάζομαι πάνω στην δομή αυτή καθ' αυτή της έκθεσης και μόλις θα έχουμε καταλήξει στη δομή θα συγκαλέσω συνάντηση και με τον σκιώδη συγητή για να αρχίσουμε να διαρθρώνουμε και να οργανώνουμε τις διάφορες ιδέες, τις πολύ σημαντικές δηλαδή ιδέες για να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των πολιτών με τον πιο αποτελεσματικά δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχουμε το χρονοδιάγραμμα, δεν το συζητήσαμε εκτεταμένα. Καλό θα είναι να έχουμε ευελιξία για το χρονοδιάγραμμα, γιατί ε, η δουλειά αυτή είναι σημαντική. Συνεργάζεστε στενά και με, τους, με τις άλλες επιτροπές. Σχέδιο έκθεσης 19 Μαρτίου, καταληκτική προθεσμία υποβολής τροπολογιών μέσα Απριλίου, ε, συζήτηση τροπολογιών το Μάιο στην Επιτροπή μας, ψήφιση στην Επιτροπή μας τον Ιούνιο και έγκριση το Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι εσείς θα κρίνετε ποια είναι τα βασικά στοιχεία που θα προέλθουν από τις άλλες επιτροπές και που θα πρέπει να μπουν στην έκθεση αυτή. Είστε απόλυτα ικανοί να ε, διεξάγετε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις με τις άλλες επιτροπές. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η έκθεση της Κριστιαν Μποσόε. Ε, ε, για την απαλλαγή 2010 Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε και τους πιο εισηγητές, κύριο Σβάρ, κυρία Χέντε, κύριε Ρούλε και οποιοδήποτε άλλος θέλει να συμβάλλει στη συζήτηση, ο κύριος Ντεγιόν και Ναδιό. Ε, δίνω το λόγο, έχει το λόγο Κρίστιαν Σίλβιο Μποζόη. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν νομίζω. Κρίστιαν παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να είμαι σύντομος. Έχω ήδη παρουσιάσει τις ιδέες μου στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό το Δεκέμβριο. Θα προσπαθήσω να κάνω μια επισκόπηση και να δώσω στη συνέχεια το λόγο στους όδης εισηγητές. <clears throat> να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληροφόρηση που μας έδωσε. Ήταν πολύ χρήσιμη. Ε, για τη σύνταξη αυτού του σχεδίου έκθεσης. Ποσοστό εκτέλεσης για τις ε, πιστώσεις ε, πληρωμών υπό τον τίτλο 12 του προπολογισμού. Αυτό έχει αυξηθεί και χαίρομαι γι' αυτό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια της προηγούμενης χρήσης. Παρ' όλα αυτά παραμένει χαμηλό σε επίπεδο πολιτικής για τους καταναλωτές. Αυτό φαίνεται στους λογαριασμούς της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ. Οι πολιτικές για τον ε, καταναλωτή δείχνουν το μικρότερο ποσοστό ε, εκτέλεσης. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να βελτιωθούν όλες αυτές οι προβλέψεις. Και θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μάθουμε γιατί είχαμε τόσο ε, χαμηλή εκτέλεση ως προς την πολιτική για τους καταναλωτές. Χαίρομαι διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναμορφώσει την πύλη, τη διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίδονται περισσότερες πληροφορίες. Θέλω να ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειές της στον τομέα αυτό και σε κάθε περίπτωση εκ μέρους όλων ημών μπορείτε να βασιστείτε στην πλήρη στηρίξη της δικής μας Επιτροπής. Το ίδιο ισχύει και για την ε, προώθηση εναλλακτικών μέσων επίλυσης προβλημάτων όπως το Solvit ή το EU Pilot. Το Solvit βεβαίως ακόμα πάσχει από την έλλειψη γνώσης από πλευράς Ευρωπαίων πολιτών και εκεί πρέπει να κάνει περισσότερη δουλειά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρόλο που και τα κράτη-μέλη και η τοπική αυτοδιοίκηση, οι εθνικές κυβερνήσεις οφείλουν να συνεργαστούν. Και βεβαίως όλοι εμείς, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα μέλη της δικής μας Επιτροπής. Νομίζω ότι το δίκτυο, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Πληροφόρησης του Καταναλωτή είναι εξαιρετικά χρήσιμο, πρέπει να το στηρίξουμε λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα, τα πορίσματα της μελέτης που παρουσιάστηκε πέρσι για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του δικτύου αυτού και για να το μάθουν καλύτερα οι καταναλωτές. Και τέλος, στο σχέδιο έκθεσης που έχω συντάξει, έχω συμπεριλάβει δύο παρατηρήσεις για τα τελωνία. Στην έκθεσή του, το ελεγκτικό συνέδριο επισημαίνει μία σειρά παρατυπιών στους, στις εθνικές δηλώσεις ως προς την ε, συλλογή των ίδιων πόρων, ε, εσφαλμένη εφαρμογή συντελεστών ε, στους δασμούς κτλ. Θα πρέπει η Επιτροπή να ασκήσει περισσότερη πίεση στα κράτη-μέλη να επιτηρήσουν πιο στενά τα τελωνία για να βελτιωθεί το θέμα με τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους. Και βεβαίως η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη παρά την καθυστέρησή της. Είναι περίπλοκο το εγχείρημα αυτό και γι' αυτό ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη της τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για τον εξυγχρονισμό των τελωνίων και να έχει πιο ρεαλιστικές προθεσμίες ως προς τη διαδικασία εφαρμογής και υλοποίησης όλων αυτών των κειμένων. Είμαι έτοιμος βεβαίως να συζητήσω μαζί σας όλα αυτά τα θέματα και με μεγάλη χαρά θα δεχθώ τα σχόλιά σας, ε, τις υποδείξεις σας και τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, και εμείς σας ευχαριστούμε. Καταφέρετε <clears throat> να συμπεριλάβατε τεράστιο υλικό τεκμηρίωσης μέσα σε μία σύντομη έκθεση. Αυτό είναι πολύ καλό. Ο κύριος Φάβε θα πάρει το λόγο και μετά η κυρία Χέντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι αρκετά σύντομος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μου ε, για τη δουλειά που έχει κάνει. Αυτά που αναφέρονται εδώ ε, μας βρίσκουν σύμφωνους. Υποστηρίζουμε τις ε, θέσεις που αναφέρονται εκεί. Πιστεύουμε ότι τα κέντρα ε, καταναλωτή έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο μέχρι τώρα για τους καταναλωτές. Θα πρέπει να συνεχίσουν και να ενδύνουν το ρόλο αυτό. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό και το κομμάτι που ονομάζουμε Better Regulation, καλύτερη νομοθεσία και για το οποίο θα πρέπει επίσης να διατεθούν α, κάποια κονδύλια στο προπολογισμό. Ε, όσον αφορά τις τροπολογίες υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος, δύο τροπολογίες από πλευρά μας, ε, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ. Και εμεί θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπουφσόη για τη δουλειά του. Μπορούμε να δεχθούμε την πρόταση που μας υποβάλλει και μπορούμε επίσης να δεχθούμε και τις τροπολογίες αυτές. Ε, είχαμε μια πολύ σημαντική συζήτηση προηγουμένως και είναι πραγματικά η ώρα να προβληματιστούμε για όλα αυτά τα θέματα. να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να βοηθήσουμε τους καταναλωτές. Δίδεται τεράστια σημασία στο Solvit. Είναι μια πολύ καλή πρόταση να έχει τη δική του ε, δημοσιονομική γραμμή, το Solvit. Και βεβαίως από εκεί και πέρα η διαδικτυακή πύλη είναι κάτι το εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ε, λειτουργεί σε όλες τις γλώσσες. Εγώ Έχω αποκτήσει πρόσβαση και επανειλημμένως την έχω επισκεφθεί, τη συστήνω ανεπιφύλακτα στους καταναλωτές. Ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε ε, ακόμα περισσότερο αυτή την ε, ηλεκτρονική πύλη η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική. Ως προς το ποσοστό εκτέλεσης ε, του προϋπολογισμού για την πολιτική για τους καταναλωτές, ελπίζω βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει τα απαραίτητα μέτρα και να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Βεβαίως, ε, όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν πριν από τις 31 Ιανουαρίου, αλλά σε κάθε περίπτωση ευχαριστούμε τον εισηγητή ε, για τη συμβολή του. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, θέλει κάποιος άλλος το λόγο, αλλιώς ε, Κρίστια να μας κάνει μια μικρή περίληψη και να δούμε ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Σβάπ και την κυρία Άννα Ρέντ για τα πολύ ευγενικά τους λόγια και για τη στήριξη που έχουν εκφράσει. στο ECCNet, στο Europe Portal και στο Solvit. Ε, θέμα που με αγγίζει ιδιαιτέρως από τη στιγμή που εγώ στο παρελθόν έχω υπάρξει εισηγητής ε, της Επιτροπής αυτής για το Solvit και πράγματι προσπαθήσαμε να ε, το καταστήσουμε περισσότερο γνωστό, περισσότερο γνωστό στην κοινή γνώμη και να πετύχουμε ε, ανεξάρτητη δημοσιονομική γραμμή πίστοσης από τον προϋπολογισμό για το Solvit. Και βεβαίως να επαναλάβω ότι με χαρά θα δεχθώ τροπολογίες, με χαρά θα δεχθώ και άλλα σχόλια και να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι με βοήθησε, μου προσέφερε τα απαραίτητα στοιχεία και τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη αυτής της γνωμοδότησης. 31 Ιανουαρίου του 2012 είναι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Η Γραμματεία μπορεί να με βοηθήσει να μου πει πότε προβλέπεται η ψηφοφορία στις 28 Φεβρουαρίου, αν δεν απατώμε, καλώς, ναι, μου το επιβεβαιώνει η Γραμματεία. Αυτά τα έχουμε ήδη συζητήσει ε, μεταξύ των ε, ε, επικεφαλής του γραφείου μου και των μελών της Γραμματείας ε, δεν είναι ένα σχέδιο γνωμοδότησης πολύ αμφιλεγόμενο. Τη χάνει ευρεία στήριξη. Είναι αρκετή η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να δώσουμε το πράσινο φω στην αρμόδια επιτροπή για να μπορέσει και εκείνη να ολοκληρώσει την έκθεσή τη. Να ευχαριστήσω όλου και να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία για άλλη μια φορά. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ για όλη αυτή τη διαχείριση του θέματος που έχετε κάνει. Έτσι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα το ψηφίσει την έκθεσή της στις 26 Μαρτίου, κάτι το οποίο είναι πολύ καλό. Λοιπόν, ο Πρόεδρος λέει ότι ε, τελειώνουμε λίγο νωρίς σήμερα. Ευχαριστεί τους διερμηνείς, ευχαριστούμε και εμείς. Έχουμε ολοκληρώσει την εξέταση του μερίσιας διάταξης. Θα ε, το απόγευμα πάλι και εκεί θα μελετήσουμε ε, την εφαρμογή της ε, οδηγίας για την ε, θα υιοθετήσουμε την οδηγία για την καταναλωτική πίστη. Και από 4.30 μέχρι 5.30 θα έχουμε συνεδρίαση των συντονιστών για την κατάρτιση της στρατηγικής. Επομένως θα τα πούμε όλοι, θα μιλήσουμε για, τις, για το κοινό σύστημα φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ε, για την καταναλωτική πίστη. Αύριο το πρωί θα ξεκινήσουμε στις 9 ακριβώς και θα ακούσουμε τον κύριο Όλε Ζων, Δανό Υπουργό Υπεχειρήσεων και Οικονομικής Ανάπτυξης. Θα του ε, θέσουμε διάφορες ερωτήσεις. Παρακαλώ στις 9 ακριβώς να ξεκινήσουμε αύριο το πρωί. Και αύριο θα ε, ακούσουμε ε, διάφορες παρουσιάσεις για θέματα δημοσίων συμβάσεων και το απόγευμα αύριο θα ασχοληθούμε με την πρόσβαση σε ένα βασικό λογαριασμό πληρωμών. Θα υπάρξει δημόσια ακρόαση αύριο το απόγευμα. Και αύριο το πρωί θα μιλήσουμε για τις δημόσιες συμβάσεις. Αυτά προς το παρόν έχω να σας πω. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.